Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχουμε την ακρόαση την οποία όλοι περιμένουμε με αδημονία για την επανεκατάσταση. Και μια που έχουμε και καλεσμένους εδώ θα ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση που ξεκινάει σήμερα και συνεχίζεται αύριο. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τους βουλευτές εγκρίνεται και έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω πρώτα απ' όλα για το γλωσσικό καθεστώς δυστυχώς δεν έχουμε ερμηνεία σε δανέζικα, ογκρικά, μαλτέζικα και γαλλικά και κάποιες άλλες ανακοινώσεις έχω τις ε, την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών συγγνώμη το άρθρο 205 πρώτα απ' όλα ο καθορισμός ε, των ε, εισηγητών ο κύριος Πόστ ε, για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία στο άρθρο 55 και η κυρία Μίλναρ από την Άλντε παίρνει την έκθεση για το πολιτέ πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και μετά για την γνωμοδότηση κυρία Στίβενς του ECR για τη γνωμοδότηση ε, καταγραφή των ατόμων ε, εν πλώ σε επιβατικά πλοία από και προς λιμάνια της κοινότητας ε, για πλοία τα οποία φτάνουν ή αποπλέουν από λιμάνια κρατών μελών. Και τέλος ο κύριος Βιώτη για την γνωμοδότηση για τους ε, κανόνες που ισχύουν για το Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης 2016 καθώς 0282 εγκρίνεται αυτές οι στάσεις ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, συνάδελφοι, καλωσορίζω τους συναδέλφους και την εισηγητριά μας, την Μαλιμπιόρκ, στο σημείο 3 το οποίο αφορά το πλαίσιο μεταγκατάστασης, επαναγκατάστασης, με συγχωρείτε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν τις επόμενες δύο ώρες με το θέμα αυτό, την μεταφορά δηλαδή υπηκών τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας από μια τρίτη χώρα σε ένα κράτος μέλος. Και βεβαίως ειδικά η επανεγκατάσταση είναι ένα ζήτημα μαζί με τη μετεγκατάσταση το οποίο είναι από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό και η συγκήτριά μας βεβαίως, συντάσσει μια έκθεση και θα την βοηθήσετε σήμερα να δει την πρόταση της Κομισιόν στον τομέα της επανεγκατάστασης. Βεβαίως αυτό σχετίζεται όπως είπαμε με τον κανονισμό που έχει στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο επαναγκατάστασης ε, των 516 του 2014 ο οποίος τροποποιείται αυτό το οποίο λέμε το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και μέρος του δεύτερου πακέτου της ε, νομοθετικής μεταρρύθμισης. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός ε, έχει στόχο, όπως έχει πει η Κομισιόν, να υπάρχει ένα μόνιμο πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία επανεγκατάσταση σε ολόκληρη την Ένωση για υποδοχή υπηκών τρίτων χωρών και απάτριτων ατόμων στην επικράτεια των κρατών μελών για να τους αποδοθεί η διεθνής προστασία. Όμως τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα αποφασίζουν πόσοι θα επανεγκαθίστανται κάθε χρόνο και το πλαίσιο αυτό, όπως προτείνει η Κομισιόν, θα εξαρτάται από τα ετήσια σχέδια επανεγκατάστασης, όπως θα τα εγκρίνει το Συμβούλιο. Αυτή είναι η πρόταση, οπότε το πλαίσιο αυτό, από αυτή την άποψη, απλά καθορίζει τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη όταν ε, θα καθορίζουμε τις ε, χώρες, εκείνες τρίτες χώρες, από τις οποίες θα λαμβάνει η χώρα η επανεγκατάσταση. Και βεβαίως να υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες για την επιλογή και την μεταχείριση των υποψηφίων προς μετεγκατάσταση. Επίσης, ορίζει κάποια κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας και ορίζει κάποια κοινή βάση για τον αποκλεισμό υποψηφίων και τον τύπο διαδικασιών είτε τακτική είτε επιταχυμένη διαδικασία δηλαδή που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όμως ε, ήδη τα μέλη, οι βουλευτές έχουν θέσει πάρα πολλά ζητήματα όπως το ζήτημα της χρηματοδότησης το ζήτημα των κριτηρίων επιλογής το θέμα της οικογενειακής επανένωσης και βεβαίως ε, το ότι όταν κάποιος έχει απορριφθεί από ένα κράτος μέλος δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση σε κανένα άλλο κράτος μέλος. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, αλλά βεβαίως το ζήτημα της επανεκατάστασης είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κοινό σχέδιο ασύλου το οποίο όπως ξέρετε δεν λειτουργεί αρκετά καλά και η σημερινή, ακρόαση θα είναι σημαντικό τμήμα αυτής της συζήτησης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα που θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μπιόρκ. Θα κάνει μια εισαγωγή και θα μας παρουσιάσει τους ομιλητές μας. Κύριε Βιόρκα, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας γιατί είναι πολύ σημαντικό και για το δικό μου έργο αλλά και για τους συναδέλφους ε, να συγκεντρώσουν όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες για να κάνω μια τεκμηριωμένη ανάλυση. Και τώρα θα συνεχίσω στα σου ειδικά, γι' αυτό παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Ε, νιώθω μεγάλη τιμή που θα ακούσω τους εμπειρογνώμονές μας, γιατί θα με βοηθήσουν ε, να εμπλουτίσω το έργο μου στην ε, πρόταση, στην έκθεση αυτή και να εκλεπτύνω τις προτάσεις μου. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι νόμοι διάβλοι για την ε, είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασχοληθούμε με εμπεριστατωμένο τρόπο με το θέμα αυτό. Και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε δίκαιοι. Και τι σημαίνει να είμαστε δίκαιοι. Το πλαίσιο μας, ε, αυτό το ενωσιακό πλαίσιο για την εμπαρακατάσταση, θα πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς κανόνες. Και θα πρέπει και οι εθνικοί και οι διεθνείς φορείς να συνεργάζονται σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο και φυσικά να αξιοποιούμε και το έργο που έχουν επιτόπου οι διάφορες ενώσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Για να επιφέρουμε προστιθέμενη αξία με το ενωσιακό πλαίσιο θα πρέπει να βελτιώσουμε την παρούσα κατάσταση και να ε, υποδεχθούμε μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώσαμε κάποια μικρή αύξηση των προσφύγων που δεχόμαστε, αλλά δεν αρκεί αυτή. Το πρόγραμμα επαναγκατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι, ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη που έχουν αναλάβει τις ευθύνε του, αλλά δεν αρκεί να αναλαμβάνουν μόνο μερικά κράτη τι ευθύνε του. Χρειάζεται αλληλεγγύη και επιμερισμός των ευθυνών. Επίσης, ε, θα πρέπει να στηριζόμαστε στις αρχές ενός ανθρωπιστικού προγράμματο που θα εξασφαλίζει προστασία σε μεγάλο αριθμό ε, προσφύγων. και θα πρέπει να δούμε αν θα επιλέξουμε το εθνικό ή το διεθνές επίπεδο. Και δεν ξέρω αν ένα τέτοιο νοσιακό πλαίσιο θα αποτρέψει τις αυθόρμητες εισόδους ή θα τις ελέγξει κάπως. Αλλά υπάρχει κίνδυνο να τα μετρέψουμε όλα αυτά σε έλεγχο μετανάστευσης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να διευκρινίσουμε όλες αυτές τις έννοιες και τους ορισμούς. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα στηρίζει τα εθνικά προγράμματα και Δεν ξέρω αν έχει νόημα να καταργήσουμε τις ε, εθνικές δυνατότητες. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να τις καταργήσουμε, θα πρέπει απλώς να τις στηρίξουμε και να τις ενισχύσουμε. Για να βελτιώσουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα από πολλές πτυχές και να έχουμε διαβουλεύσεις ε, με ενδιαφερομένους ε, διεθνείς και εθνικούς εμπειρογνώμονες, εθελοντές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και γι' αυτό οι καλεσμένοι μας θα μας παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρία και τη δική τους γνώμη για να μην κάνουμε λάθος στην πορεία που θα χαράξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Έχουμε το EMN, e το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Μετανάστευση, που θα μα παρουσιάσει μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των προγραμμάτων επανεγκατάσταση των κρατών μελών, πολύ σημαντική μελέτη. Επίση, θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη ΥΠΑ των Ηνωμένων που είναι ο κεντρικό ε, παράγων ε, σε θέματα αυτά. Επίσης ε, θα ε, ακούσουμε εκπροσώπους ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και θελοντικών οργανώσεων που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των προγραμμάτων εμπενεγκατάστασης Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Όσκαρ Εκμπλατ που θα μας παρουσιάσει την άποψη της, του Σουηδικού Οργανισμού Μετανάστευσης και του Εθνικού Προγράμματος Επανεγκατάστασης της Σουηδίας και έχουμε και τον κύριο Πατρίς Κεσάντα από την IOM, τη Διεθνή Οργάνωση για τη Μετανάστευση. Χαίρομαι πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να ακούσω τις παρουσιάσεις σας. Ευχαριστούμε κυρία Πιόρκ, έχετε απόλυτο δίκιο και αφού ακούσουμε τους ε, εμπειρογνώμονές μας θα ξαναδώσουμε το λόγο στην ε, εισηγήτρια για πιο επιμέρους ερωτήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την παρουσίαση της μελέτης για την επανεγκατάσταση που προβλέπει συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων επανεγκατάστασης των κρατών μελών. Ε, θα μας την παρουσιάσει ο κύριος Ρουσέλ από την Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα και τον κύριο και την κυρία Μπιόρκ και τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που με κάλεσαν και μου δίνουν την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την ολοκένουργια μελέτη για το θέμα αυτό, Εκφράζω τη χαρά μου για την παρουσία μου εδώ. Όταν αρχίσαμε να εκπονούμε τη μελέτη πριν από ένα χρόνο, ελπίζαμε ότι θα προκαλούσε κάποιο ενδιαφέρον, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα ενταχθεί άμεσα στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ελπίζω όσοι τη διαβάσουν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούν τα προγράμματα επανεκατάστασης και ανθρωπιστικής εισδοχής στα διάφορα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το υπόβαθρο αυτής της μελέτης. Όπως γνωρίζετε, είχαμε αυξανόμενο ρυθμό προσφύγων παγκοσμίω και η κατάσταση των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μάλλον χαοτική. Είχαμε έντονες μεταναστευτικές πιέσεις και οι πρόσφυγες διαλέγουν ε, παράτυπους διάβλους και επικίνδυνα ταξίδια για να φτάσουν στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα και πιο νόμιμα ε, μονοπάτια, νόμιμους διάβλους ε, εισόδου και η επανεγκατάσταση είναι ένας τέτοιος νομικός νόμιμος διάβλος. Ε, θα πρέπει λοιπόν να το, να το βελτιώσουμε και να το διαβρύνουμε καλύψαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 23 κρατημέλη και την Ορβηγία για να δούμε πώς λειτουργούν τα προγράμματα επανεγκατάστασης. Εξετάσαμε κάποιες νέες ε, εξελίξεις. Ε, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και να αντιλήσουμε και κάποια διδάγματα. Επίσης, ε, εξετάσαμε κάποια προγράμματα ιδιωτικής χορηγίας που εφαρμόζονται σε κάποια κράτη-μέλη. σας παραπέμπω στην έκθεση. Υπάρχουν τρία διαφορετικά format. Φυσικά έγινε μια ανάλυση της κατάστασης και των πολιτικών των κρατών μελών. 61 σελίδες κρατάει αυτή η ανάλυση. Και επίσης, ε, για όσους δεν έχουν το χρόνο να διαβάσουν την πλήρη μελέτη, υπάρχει μια σύνοψη οκτασέλιδη ε, με τα βασικότερα πορίσματα και Τέτοιου είδου εκθέσει στηρίζονται σε εθνικέ εκθέσει με τη συμμετοχή κρατών μελών. Έχουμε και τι 24 λοιπόν εθνικές εκθέσεις για τα προγράμματα επανεγκατάσταση που επίση ε, μπορούμε να σα παράσχουμε για μελέτη. Η μελέτη μα καλύπτει 23 κράτη-μέλη και την Ορβηγία. Δεν καλύπτονται η Δανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ελλάδα. Θα ήθελα να σα πω εν συντομία πώ ορίζουμε του διάφορου όρου Καταρχήν Επανεγκατάσταση είναι η μεταφορά ενό υπηκοτρή χώρα ή Απάτριδο, ε, κατά αίτημα τη υπερσαρμοστία και με βάση την ανάγκη διεθνού προστασία, από μια τρίτη χώρα σε ένα κρατος όπου επιτρέπεται να παραμείνει ως ε, με το καθεστώ του πρόσφυγα ή παρόμοιο καθεστώς. Τώρα, ε, η παρομοιο καθεστω τωρα η εννοια τη ανθρωπιστική εισδοχή δεν έχει συγκεκριμένο ορισμό, αλλά για τα πλαίσια τη μελέτη θεωρούμε παραφέρει με την επανεγκατάσταση αλλά δεν, δεν είναι πανομοιότυπος ορισμός. Μπορεί να έχουμε ένα τχόκ σύστημα για σύντομη περίοδο ή για συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει συνήθως αυτό, αυτή η έννοια μακροπρόθεσμη προοπτική. Και να σας δώσω μία σύντομη απεικόνηση των στατιστικών στοιχείων που έχουμε. Κατά την πενταετία 2011-2015, οι βασικέ χώρε επανεγκατάσταση, οι βασικέ χώρε υποδοχή ήταν Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια Ολλανδία, Γαλλία και Αυστρία. Και πολλέ άλλε χώρε που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν ξεκινήσει συστήματα επανεγκατάσταση, προγράμματα επανεγκατάσταση, αλλά με πολύ χαμηλά νούμερα. Έχουμε και μια άλλη γραφική παράσταση που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για να αντιληφθεί και το υπόβαθρο της επαναγκατάστασης, συγκρίναμε τον αριθμό των τόπων που έχουν επαναγκατασταθεί μετά από και τις θετικέ αποφάσεις για χορήγηση άσυλο. Δηλαδή, η, η γαλάζια στήλη δείχνει αυτούς που έχουν λάβει θετική απόφαση για την αίτηση ασύλου γιατί η χορήγηση ασύλου είναι ο βασικός τρόπος παροχής προστασίας, διεθνούς προστασίας. Ε, αλλά αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τον ελάχιστο αριθμό των αιτήσεων και των αποφάσεων για επανεγκατάσταση και ε, ανθρωπιστική εισδοχή. Βλέπετε ότι κάποιες χώρες έχουν επαναγκαταστήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρόσφυγες, έχουν μακροχρόνια πείρα. Αλλά από το 2010 και μετά ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα επανεγκατάσταση έχει αυξηθεί. Και ιδιαίτερα την τελευταία διετία, 2015-2016, εκτοξεύτηκε στα ύψη ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα επανεγκατάστασης. Εδώ μπορούμε να ομοδοποιήσουμε τι χώρε μέλη σε τέσσερι ομάδε. Έχουμε καταρχήν τι ε, χώρε που έχουν μόνιμα προγράμματα επανεγκατάσταση. Έχουμε τη δεύτερη ομάδα χωρών που έχουν προγράμματα και επανεγκατάσταση και πιο ad hoc προγράμματα ανθρωπιστική εισδοχή, Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε κάποιε χώρε που έχουν ε, ad hoc ε, προγράμματα επανεγκατάσταση και ανθρωπιστικής ε, εισδοχή, αλλά όχι μακροχρόνια προγράμματα επανεγκατάσταση. Και τελευταία ομάδα είναι των χωρών που τώρα αρχίζουν και καταρτίζουν προγράμματα επανεγκατάσταση. Κύπρος, Κροατία, Λιθουανία, Λετωνία και Μάλτα είναι οι χώρες της τελευταίας ομάδας. Η βασική σύγκριση μεταξύ των χωρών τώρα. 17 χώρε μέλη και η Νορβηγία έχουν ήδη προγράμματα επανεγκατάστασης ή ανθρωπιστικής εισδοχής, είτε είχαν στο παρελθόν, ενώ έξι χώρες μέλη δεν είχαν ουδέποτε μέχρι στιγμής εμπειρία με επανεγκατάσταση ή ανθρωπιστική εισδοχή. Και ενώ τα, οι βασικοί στόχοι των κρατών μελών και των προγραμμάτων του είναι παρόμοιοι, δηλαδή η παροχή προστασίας ε, στου χρήζοντε βοήθεια, βοήθεια στι χώρε πρώτη περίθαλψης, ανέβρεση βιώσιμων λύσεων, τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επανεκατάσταση διαφέρουν μεταξύ του. Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα και μηχανισμοί, μερικέ χώρε χρησιμοποιούν ποσοστώσεις, υπάρχουν διαφορετικέ προτεραιότητε επιλογή, αλλά και διαφορετικέ μέθοδοι επανεγκατάσταση. Και θα ήθελα εν συντομία να σας αναλύσω και αυτά τα σημεία. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους ε, επιλογής και το καθεστώς των δικαιούχων, η Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών ε, εντοπίζει, ε, ε ταυτοποιεί ε, και αναγνωρίζει υποψηφίου για επανεγκατάσταση, αλλά την τελική απόφαση για το κατά πόσο θα λάβει η χώρα μια τέτοια επανεγκατάσταση τη λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Και γενικώ ε, αυτό γίνεται με τη χρήση τη ε, της μεθόδου που στηρίζονται στους φακέλους, στα ντοσιέ. Και αυτό το κάνουν οι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη, μετά τα στοιχεία που τους υποβάλλει η πατιαρμοστία. Γενικώ ε, η επαναγκατάσταση προϋποθέτει αναγνώριση του καθεστώτος ε, πρόσφυγα από την υπατερμιστία ε, πριν την εισδοχή. Και μερικά κράτη-μέλη δέχονται δικαιούχους και επικουρική προστασίας, ενώ μερικέ επαναξιολογούν την προστασία, την, αναγνώριση προστασίας που έχει κάνει η πατιαρμοστή, ενώ άλλε στηρίζονται στην αναγνώριση και την παραπομπή του, της η ανθρωπιστική ζωή μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση ε, από την υπατερμοστία και έχει προσωρινό χαρακτήρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια προτεραιότητα και επιλογή. Μερικά κρατημέρια χρησιμοποιούν επιπλέον κριτήρια, είδο και βαθμός τροτότητα, για παράδειγμα, επιζήσαντε από βασανιστήρια ή βία ή χρήζοντε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το θέμα της ηλικία, ε, ηλικιωμένοι οι παιδιά, οι μητέρες ε, μόνες τους. Ε, μερικοί λαμβάνουν υπόψη την οικογενειακή ενότητα, προηγούμενους δεσμούς συγκεκριμένου πρόσφυγα με τη χώρα προορισμού και κάποιες χώρες επίσης κάνουν και μία εκτίμηση του δυναμικού ένταξη που έχει ο συγκεκριμένος πρόσφυγας. Επίσης, ε, κριτήρια αποκλεισμού ή κατάρριση των προτεραιοτήτων ε, που χρησιμοποιουνται απο από μερικά κράτη-μέλη. Και κάποια κράτη έχουν και έκτακτες ποσοστώσεις στα πλαίσια της συνολικής ποσόστοσης επανεγκατάστασης για να επανακαταστήσουν ε, έκτακτες περιπτώσεις. Τρεις χώρες, Ολλανδία, Σουηδία και Φιλανδία έχουν τέτοιε έκτακτε ποσοστώσει. Ό,τι αφορά το καθεστώ που αναγνωρίζεται, ποσοστώσει και γεωγραφικέ προτεραιότητε, οι περισσότερες χώρες μέλη χορηγούν όσου ε, ε, όσους έρχονται ως ετούντε ετούντες προστασία, το καθεστώς του πρόσφυγα ή ε, δικαιούχου προστασίας, αλλά οι διατάξεις για την στέγαση και τις ρυθμίσεις ένταξης ποικίλουν. Ε, χώρε χώρες, περισσότερες έχουν αιτήσει ή ποσοστό για την επαναγκατάσταση, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν γεωγραφικέ προτεραιότητε και εστιάζονται κυρίω στου Ήρου πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση μετά την άφηξη στα κράτη-μέλη, μερικά κράτη-μέλη ε, ε, στεγάζουν τους ε, επαναγκαταστημένου πρόσφυγες σε κέντρα υποδοχή ή ε, διέλευση, ενώ άλλοι, άλλα κράτη-μέλη προβλέπουν αμέσω μόνιμη ε, στέγαση. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών στο τι προσφέρουν ε, στους πρόσφυγες ό,τι αφορά τα, ε, κάποια επιδόματα, μαθήματα, εκμάθηση γλώσσας ή πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης, κάποια κρατημέλη έχουν εσωτερικό μηχανισμό κατανομής μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, δήμων ή περιφερειών, αλλά δεν ισχύει για όλα τα κρατη Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική χορηγία. Και εδώ έχουμε κάποιες διαφορές, γιατί εδώ έχουμε συμμετοχή και ιδιαιτών. Μόνο πέντε χώρες μέλη όμως έχουν ε, επίσημα προγράμματα ιδιωτικής χορηγίας. πολύ μικρή είναι σχετική αριθμή, με εξαίρεση τη Γερμανία, ε, που οι περισσότεροι έχουν ε, ε, επανακατασταθεί με βάση την οικογενειακή επανένωση. Βέβαια, η, η ιδιωτική χορηγία ε, είναι ευρύτερη από την οικογενειακή επανένωση και καλύπτει ευρύτερου οικογενειακού δεσμού. Μάλιστα, τέτοιου είδου προγράμματα έχουν μερικέ φορέ και κάποια θρησκευτική διάσταση, επικεντρώνονται σε θρησκευτικέ ομάδε. Πάντω, ε, η εμπειρία για τέτοια προγράμματα ιδιωτική χορηγία είναι περιορισμένη. Αν και μερικέ χώρε έδειξαν ενδιαφέρον. Τώρα, να σα ε, πω δύο λόγια για τι προκλήσει που εντοπίσαμε. Μπορούν να διαχωριστούν σε προκλήσεις πριν την ε, αναχώρηση και μετά την άφηξη. Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση, ε, μακροχρόνια διαδικασίες επιλογής, καθυστερημένες μεταφορές, ε, εμπόδια επιμελητιακά, κίνδυνη ασφάλειας, αδυναμία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, η παροχή πληροφοριών πριν την αναχώρηση και προσανατολισμός και αυτό είναι σημαντική πρόκληση γιατί χρειάζονται πόροι, χρειάζεται προσωπικό για να εξασφαλίσει αυτή την ενημέρωση και είναι δύσκολο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ή να ενημερωθούν επαρκώς οι υποψήφοι για επανεγκατάσταση για το τι, τι πρέπει να περιμένουν όταν φτάσουν. Σε ό,τι αφορά την άφηξη και την περίοδο μετά την άφηξη, ε, η εξασφάλιση στέγης, δεν υπάρχουν αρκετές κατοικίες, η οργάνωση εκμάθησης της γλώσσας, η παροχή δικής προστασίας και η εξασφάλιση εργασιακών ευκαιριών. Τώρα, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις. Χρειάζεται καλό συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών καταρχήν. Αυτό έδειξε η εμπειρία μας μεταξύ του εθνικού και του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου. Πρέπει να παρέχονται επαρκείς και ρεαλιστικές πληροφορίες και σωστός πολιτιστικός προσανατολισμός για να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι και να γίνει σωστή διαχείριση των προσδοκιών τους. Να γνωρίζουν δηλαδή οι άνθρωποι τι να περιμένουν όταν φτάσουν στη χώρα υποδοχής. Πρέπει να βελτιωθεί και η παροχή στέγης στη χώρα προορισμού και η παροχή μόνιμης στέγης αμέσως μετά την άφηξη του πρόσφυγα. Και μια άλλη πρόκληση είναι η διεύρυνση του ρόλου των τοπικών κοινότητων και των εθελοντών, ώστε να μην εγκαταλείπονται στη μοίρα τους μετά την άφεξή τους οι πρόσφυγες. Μερικές χώρες μάλιστα έχουν και πρωτοβουλίες όπου άλλοι πρόσφυγες που ήδη έχουν επανεγκατασταθεί προσφέρουν βοήθεια και στήριξη στους νεοαφιχθέντες. Γενικά συμπεράσματα. Οι δεσμεύσεις και υποσχέσεις ε, που έχουν κάνει οι χώρες έχουν αυξηθεί αισθητά για την επανεγκατάσταση τα τελευταία χρόνια, αν και το, το ποσοστό της επανεγκατάστασης εξακολουθεί να είναι χαμηλό και εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό για να θεωρηθεί ως αποτελεσματική εναλλακτική στην παράτυπη ε, είσοδο Και για να αποτελέσει επανεγκατάσταση πραγματική εναλλακτική λύση θα πρέπει να αξιθούν οι αριθμοί επανεγκατάσταση. Θα πρέπει να προωθηθεί η επανεγκατάσταση ω συνταγμένη διαδικασία με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και την ανάδειξη των τοπικών και θετικών εμπειριών. Θα πρέπει ε, να προαγάγουμε τι ευκαιρίε που προσφέρει η επανεγκατάσταση και για τους τοπικού ε, πληθυσμού που υποδέχονται του πρόσφυγες ε, και τι προγραμματισμό χρειάζεται για κάτι τέτοιο. Και ένα άλλο σημείο ίσω ήταν ε, η αξιοποίηση αυτών των προγραμμάτων ιδιωτική χορηγία. Χώρε όπω ο Καναδά χρησιμοποιούν τέτοια ιδιωτικά προγράμματα πολύ σε, μεγαλύτερο βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμεί να διευρύνουμε περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα. Για να την διερευνήσουμε πρώτα. Αυτά ευχαριστώ και όσοι έχετε περαιτέρω απορίες μπορείτε να με μου στείλετε για να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατάλαβα είναι όλα διαθέσιμα και διαδικτυακά, οπότε μπορείτε να τα δείτε και να δείτε και αναλυτικά στοιχεία για την ανάλυση. Εσείς βέβαια μας παρουσιάσετε την ευρύτερη εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ και φυσικά θα ακούσουμε ερωτήσει στο τέλο ε, μετά από όλε τι παρουσιάσει. Αν υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο φλέγεστε να ρωτήσετε, παρακαλώ να μου το πείτε, ιδίω αν πρέπει να φύγετε νωρίτερα ή υπάρχει κάποιο άλλο λόγο ε, Να μου το πείτε, να σα δώσω το λόγο. Αλλιώ, θα ακούσουμε όλε τι ερωτήσει στο τέλο. Τώρα έχουμε την αξιολόγηση τη ΥΠΑ τη για του πρόσφαγε για την πρόσταση. Έχουμε εδώ τον Μάντα Τζι Σεντράκ, ο οποίο είναι ο ε, ανώτερος υπάλληλο έχει σε θέματα επανεγκατάστασης ε, της υπατουσαρμορτίας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Επιτροπή που μας ε, δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό επίσης να δούμε εδώ και τα μέλη του πάνελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε την ουσία της επανεγκατάστασης. Πρόκειται ε, για μια διαδικασία η οποία ε, εκφύσεως είναι ε, μια διαδικασία συνεργασίας και εδώ λοιπόν έχουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, φορείς οι οποίοι πραγματικά υλοποιούν τα θέματα της επανεγκατάστασης. Θεωρούμε ότι η ευκαιρία αυτή είναι μία εκ των πολλών, ίσως μία από τις πρώτες ας πούμε επίσημες ευκαιρίες ε, για να ε, συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα προκειμένου να δούμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό πλαίσιο. Επίσης ε, θα θέλαμε επί τη ευκαιρία όχι μόνο να σας παρουσιάσουμε τις αρχικές μας σκέψεις για το πλαίσιο αυτό, αλλά και να ακούσουμε και να συζητήσουμε από κοινού διότι θεωρούμε ότι αυτό εν τέλει θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα εύρωστο και βιώσιμο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανεγκατάσταση, το οποίο άλλωστε ε, επιθυμούμε. Και βεβαίως ε, αυτό ε, θα είναι και μια ευκαιρία να σας πούμε εμείς τη δική μας τη θέση, που ελπίζουμε να τη μοιραστείτε με τα κράτη-μέλη ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα στις επόμενες ημέρες. Επιτρέψτε μου λοιπόν καταρχάς να σας πω ότι το πλαίσιο είναι προφανώς ευπρόσδεκτη συνεισφορά ε, στον καταμερισμό των βαρών και πολύ επίκαιρη. Δεν χρειάζεται τώρα να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συμβαίνει επιτέπου ε, και το γεγονός ότι υπάρχει μια παγκόσμια διαδικασία εκτοπισμού. Η εκτιμά ότι το 2017 θα έχουμε τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια άτομα τα οποία θα χρειάζονται επανεγκατάσταση. Επομένως, είναι πάρα πολύ επίκαιρο το πλαίσιο υπ' αυτήν την έννοια και ε, παρουσιάζει κάποια πολύ σημαντικά βήματα ώστε να καταλήξουμε σε ένα ε, πιο εύρωστο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανεγκατάστασης και φυσικά συνεισφέρει και στις ε, παγκόσμιο καταμερισμό των βαρών. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει συνέπεια με τα όσα δεσμεύτηκαν να κάνουν τα κράτη-μέλη στη δήλωση της Νέας Υόρκης ε, της 19ης Σεπτεμβρίου. Γίνεται έκκληση για επέκταση της επανεγκατάστασης και αναζήτηση άλλων οδών για την υποδοχή των προσφύγων. Η ύπατη αρμοστία λοιπόν καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία νομίζω ότι είναι καρπός ε, πολύ μεγάλης συνεργασίας και φυσικά και ε, την υποστηρίζει και η πατεραρμοστία και ε, οι υπόλοιπε οργανώσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις εταιρικές σχέσεις οι οποίες διέπουν την επανεγκατάσταση από ε, τότε που ξεκίνησε. Η ύπατη στα πλαίσια της επανεγκατάστασης στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, προσπαθεί να αναπτύξει ένα πολύ ε, εύρωστο πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουμε συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουλίου του 2015 αποτέλεσε πολύ σημαντικό ορόσημο Είχαμε ε, ένα πολύ μεγάλο ρυθμό, περίπου 11 ε, χώρες ε, οι οποίες ξεκίνησαν διαδικασίες επανακατάστασης μέσω αυτού του προγράμματος για πρώτη φορά. Επομένως, αυτό το πνεύμα εταιρικής σύμπραξης και συνεργασίας θέλει να επισημάνει η Πατιαρμοστία στη συνέχεια. Και ο ρόλος ο δικός μας ποιος είναι. Θεωρούμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε, μεν, αλλά μπορούμε επίσης και να ε, προσφέρουμε την προστιθέμενη αξία μας ε, στην όλη διαδικασία. Θα θέλαμε το πλαίσιο αυτό να ευθυγραμμιστεί με τις ε, υπάρχουσες αρχιτεκτονικές δομές. Πρόκειται για ένα πλαίσιο το οποίο διέπει τις διαδικασίες επανεγκατάστασης με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένως, θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. That would be of interest to ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να θέξω μεταξύ άλλων είναι καταρχάς ότι χαιρόμαστε που στο πλαίσιο αναφέρεται η πρόθεση να ε, συμπληρώσει το πλαίσιο το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας και επανεκατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης για τον πλούτο της εμπειρίας που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα επανεκατάστασης. Το θέμα αυτό λοιπόν του, της συμπληρωματικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα μας επιτρέψει να προσθέσουμε στοιχεία στα υπάρχοντα εθνικά προγράμματα. Δεν θα υποκαταστήσει τα εθνικά προγράμματα, αλλά θα προσφέρει περισσότερα πάνω των, άνω των ε, εθνικών προγραμμάτων. Και φυσικά κάτι το οποίο είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές καλές πρακτικές στα εθνικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα ή ποσοστό εκτάκτου ανάγκη και κάποιες άλλες πρακτικές στα εθνικά προγράμματα, τα οποία πρέπει να συνεχίσουν προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν αυτό που αποκαλούμε εμεί ε, ε, ε, επιτόπιες λύσει για να καλύψουν πολύ συγκεκριμένε ανάγκες. Ε, το πλαίσιο λοιπόν υποκαθιστά, ε, εάν μάλλον το πλαίσιο υποκαθιστούσε τα εθνικά προγράμματα, θα χάναμε αυτές τις ευκαιρίες. Το σκεπτικό είναι να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά και θα ακούσουμε μετά από τον Όσκαρ από τη Σουηδία ότι πρόκειται για ένα από τα προγράμματα τα οποία ε, μπόρεσε να καλύψει και αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες και θα θέλαμε να δούμε να, κάποιες από αυτές τις εμπειρίες να τις εκμεταλλευτούμε και να προχωρήσουμε βάσει αυτά. Θα θέλαμε λοιπόν το πλαίσιο να συνεισφέρει και σε μεγάλο αριθμό ατόμων που επανεγκαθίσταται. Ακούσαμε ότι οι ανάγκες είναι πολύ ψηλές, επομένως χρειαζόμαστε ε, αριθμό ατόμων που να είναι αντίστοιχο των αναγκών. Και επίσης θα μας ενδιαφέρει και η οικονομική αλλά και η τεχνική και θέλω να τονίσω ότι την τεχνική πτυχή. Θα παρασχεθεί τεχνική βοήθεια σε χώρες οι οποίες δεν έχουν μακρά εμπειρία εφαρμογής επανεγκατάστασης όσον αφορά τη δυνατότητα πρόβλεψης και σχεδιασμού. Ξέρουμε ότι το πλαίσιο ως στόχο έχει να ε, υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών μελών. Ε, κράτη ε, τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα με την ύπατη αρμοστία εδώ και χρόνια γνωρίζουν την αξία του σχεδιασμού και της πρόβλεψης σε θέματα επανεγκατάστασης. Το γεγονός λοιπόν ότι θα υπάρχει ένα προβλέψιμο πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα επανεγκατάστασης για την επόμενη χρονιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα θέλαμε βέβαια ο σχεδιασμός αυτό στο μέτρο του, δυνατών, του δυνατού να ευθυγραμμιστεί με τα ε, προγράμματα της ΥΠΑ της Αρμοστίας για επανεγκατάσταση, η οποία, ε, ε όπως γνωρίζετε, βασίζεται στην ετήσια τριμερή διαβούλευση για την επανεγκατάσταση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο. Υπάρχει επίσης περιθώριο όχι μόνο για ε, ένα κύκλο ετήσιο σχεδιασμού και μία ετήσια προσέγγιση, αλλά να επικεντρωθούμε και σε ένα πολιετές ε, ε, σχέδιο και σε πολιετή διαδικασία επανεγκατάστασης. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε κάποιες περιοχές. Η πρόταση αναφέρεται σε μια δυτή διαδικασία, τη συνήθι διαδικασία και την ταχεία διαδικασία. Και επίσης ε, τονίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρώνει τη διαδικασία όσο το δυνατόν συντομότερα. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η λύση και θεωρούμε ότι ο τρόπος να το επιτύχουμε σημαίνει ότι και η Πατιαρμοστία και όλες οι χώρες που συμμετέχουν στην επανεγκατάσταση θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις ε, και ε, θα βλέπουμε και τι έρχεται να προσθέσει ο καθένα στη διαδικασία. Πρόκειται για κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει η Πατιαρμοστία εδώ και αρκετό καιρό με κάποιες χώρες. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ ευπρόσδεκτο αυτό το στοιχείο. Κάτι άλλο το οποίο θα θέλαμε είναι ίσως στο πλαίσιο να συμπεριληφθεί και ένας μηχανισμός ο οποίος θα επιτρέπει και επανεγκατάσταση κάποιων ατόμων λόγω κατεπίγουσας ανάγκης. Να λάβουμε λοιπόν υπόψη κάποιες θετικές εμπειρίες που υπάρχουν από τα υφιστάμινα ε, προγράμματα σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα εντάξουμε και αυτά στο πρόγραμμα. Κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να επισημάνουμε όταν συζητούμε την συνήθη διαδικασία και την ταχεία διαδικασία είναι ότι η πρόταση τα συνδέει με το καθεστώς ε, που θα ε, δίνεται σε κάποιον ε, που κάνει αίτηση. Αν είναι ταχεία διαδικασία χρειάζεται και επικουρική προστασία ενώ εάν είναι συνήθιση διαδικασία μπορεί να απλώς μετανάστευση. Η εμπειρία εφαρμογή από την Τουρκία, η πρόσφατη εμπειρία, δείχνει ότι αρκετά κρατημέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταχεία διαδικασία χωρίς να υπονομεύουν ε, τι καθεστώς ε, θα αποδοθεί στον κάθε πρόσφυγα. Επομένως πρέπει να ε, μην συγχαίουμε τα δύο εργαλεία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό και το συζητήσαμε αυτό και στο πλαίσιο τη συνήθους κυκλοφορία ατόμων στην Ευρώπη. Είδαμε, για παράδειγμα, πέρσι ότι γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις για τη μετανάστευση και τη διαχείρισή της. Η επανεγκατάσταση με την πάροδο των ετών ε, είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους πρόσφυγες και άτομα τα οποία χρήζουν ε, προστασίας μπορούν να ταξιδέψουν και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε μια νέα χώρα. Η επανεγκατάσταση μπορεί να έχει κάποια κοινά με τις ιδιαιτερότητες ε, που έχουμε στη μετανάστευση και στις διάφορες διαδρομές. Είναι στην πραγματικότητα όμως μια διαφορετική διαδρομή. Και τα βασικά στοιχεία είναι να λάβουμε υπόψη και τα θέματα της προστασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι τα κράτη-μέλη εν γέννη επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης. Η μετανάστευση από το σχεδιασμό της δεν είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Είναι ένα εργαλείο για την προστασία των προσφύγων και για την προσφορά μιας βιώσιμη λύσης ε, για τα προβλήματα των προσφύγων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση αυτή, την οποία θα θέλαμε να τονίσουμε ε, όταν εξετάζουμε συνολικά την πρόταση. Ε, εμείς είμαστε υπέρμαχοι και το έχουμε συζητήσει με αρκετές χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με την επανεγκατάσταση. Ε, το στρατηγικό χαρακτήρα της επανεγκατάστασης, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επανεγκατάσταση για να προσφέρουμε στοιχεία στους πρόσφυγες που δεν ε, τους ενδιαφέρουν όταν συζητούν αρχικά την επανεγκατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επανεγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται υπό όρους ε, ε, εάν εφαρμόζεται η συμφωνία επιστροφών ή την πρώτη χώρα υποδοχής ή την ευθύνη ή τη δράση της πρώτης χώρας στην οποία γίνεται αίτηση ασύλου για να έχουμε κυκλοφορία εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της και δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός της. Στο πλαίσιο αναλύεται το σημείο αυτό αρκετά διεξοδικά και εμείς πιστεύουμε, όπως σας είπα, η δομή και το πλαίσιο της επανεγκατάστασης, ε, το οποίο χρησιμοποιεί η Πατιαρμοστία, κάθε χρόνο πριν από την ε, τριμερή διαδικασία επανεγκατάστασης τον Ιούνιο, δημοσιεύουμε τις ε, παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης. Και το έγγραφο αυτό τονίζει σε ποιε περιοχές και σε ποιου τομεί θεωρεί η υπατερμοστή ότι θα πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση και για στρατηγικούς λόγους αλλά και ως μια βιώσιμη λύση και μια λύση για προστασία. Θεωρούμε ότι η επιλογή της περιοχής στην οποία θα πρέπει να γίνεται επανεγκατάσταση και τα στοχευμένα προγράμματα επανεγκατάσταση τα οποία αναφέρονται στο σχέδιο κανονισμού θα πρέπει ε, να γίνονται βάσει αυτού ε, του εγγράφου και τα προγράμματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούν την επανεγκατάσταση θα μπορούσαν να ε, λάβουν στοιχεία από αυτό. Γι' αυτό, για παράδειγμα, τη σήμερα ημέρα επικεντρωνόμαστε στους Σύρους. Ε, συμφωνεί και η Πατιαρμοστία γιατί οι Σύροι είναι το 40% των παγκοσμίων αναγκών επανεγκατάστασης. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε αυτό το νέο πλαίσιο με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική δομή και πλαίσιο επανεγκατάστασης. Μπορεί να επαναλαμβάνω τα ίδια εδώ, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο μέσω αυτής της ετούσιας ε, τριμερούς διαδικασίας ε, ε, διαβουλεύσεων ε, για την επανεγκατάσταση. Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά εδώ και χρόνια και μέσω αυτού μπορέσαμε να συνεργαστούμε με χώρε και άλλου ενδιαφερομένου, μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλου φορεί που ασχολούνται με θέματα επανεγκατάσταση για να καθορίσουμε μια σειρά αποδομέ που επιτρέπουν την επανεγκατάσταση τι είναι επανεγκατάσταση, ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για επανεγκατάσταση, πώς γίνεται η επανεγκατάσταση και ποιος είναι ο ρόλος και οι ευθύνες του καθενός που συμμετέχουν σε θέματα επανεγκατάστασης. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν σημαντικό το πλαίσιο το να ε, συμπληρώσει όλα αυτά και να χρησιμοποιήσει αυτά ως στοιχείο για να προχωρήσει περαιτέρω και να μην έχουμε μια παράλληλη διαδικασία που επαναλαμβάνει πράγματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πτυχή. Ε, κάτι ακόμα το οποίο θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους διαφορετικούς ρόλους και ευθύνης του καθενός στην επανεγκατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε ρητά αυτό στο πλαίσιο ίσως και να το εξηγήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διάφοροι εταίροι που συμμετέχουν στην επανεγκατάσταση ο καθένας θα κάνουν αυτό το οποίο τους ε, ε, αναλογεί. Ε, για παράδειγμα, ε, θα υπάρχει αναγνώριση στις ταυτότητες, οι χώρες θα διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη κυβερνητική προσέγγιση, ε, μπορούμε να έχουμε άλλο φορέα ο οποίο θα ασχολείται με την διαδικασία πρώτη αναχώρηση. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει μπορούν να ασχοληθούν με την αναγνώριση ταυτότητα αλλά και την υποδοχή και την ένταξη. Πρόκειται λοιπόν για ένα αμάλγαμα εταίρων που συνεργάζονται προκειμένου να καταφέρουν όλε αυτέ τι πτυχέ. Επίσης, μας επιτρέπει να ε, δούμε τους διάφορους στόχους της επανακατάστασης. Όταν αναφέρομαι σε στρατηγική χρήση επανακατάστασης, θα δείτε ότι εκφύσεως η ύπατη λόγω της εργασίας της που έχει σε διάφορες χώρες, βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να συμβουλεύσει πότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η επανακατάσταση με στρατηγικό τρόπο. Δύο λόγια πολύ σύντομα τώρα για το θέμα της επανένωσης των οικογενειών και την επανεγκατάσταση και τα κριτήρια. Βλέπουμε ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρονται σε μέλη οικογενείας ξεχωριστά και νομίζουμε ότι εάν τα αναφέρουμε έτσι, η πρόταση, χωρίς να το αντιλαμβάνεται δεν κάνει τη σωστή διάκριση μεταξύ τη δυνατότητα επανένωσης οικογενειών και επανεγκατάστασης ως μέσο προστασίας και βιώσιμη λύση για τους πρόσφυγες. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια σημαντική πτυχή την οποία θα πρέπει να επανεξετάσουμε ε, καθώς προχωρούμε και θα θέλαμε να ζητήσουμε από τις διάφορες χώρες να θεσπίσουν προγράμματα επανένωσης οικογενειών βάσει της δήλωσης της Νέας Υόρκης. Τέλος, η πρόταση αναφέρεται στην ε, Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου Επανεγκατάστασης. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια δομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορεί να προσαρμοστεί προκειμένου να καλύψει τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ολοκληρώσω και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις ε, που θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Όπως σας είπα, ε, είναι η πρώτη ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε και να τίνουμε δίκονους βεβαίως τα όσα έχετε να πείτε κι εσείς και θα σας ε, δώσουμε πολύ πιο διεξοδικά στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη γρηγόρη. Ναι, πάρα πολύ χρήσιμα αυτά γιατί υπάρχει το ζήτημα του πώς το Κοινοβούλιο θα υποποιήσει αυτή την πρόταση. Λοιπόν, η Μάλλον Πιόρκ θέλει να παρέμβει τώρα έτσι λίγο σύντομα. Ναι, σύντομα, γιατί έχουμε τρεις παρουσιάσεις ακόμα. Θα περιμένουμε βεβαίως την παρέμβασή σας, αλλά είναι ενδιαφέρουσες οι αρχικές σας παρατηρήσεις και θα ήθελα να αναπτύξετε ακριβώ το πώς δεν θα δημιουργήσουμε παράλληλες αλλά συμπληρωματικές δομές και πώς το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδεθεί με την υφιστάμενη αρχιτεκτονική με καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και οπωσδήποτε θα είμαστε σε επαφή μαζί σας. Ναι, ναι, σωστά αυτά. Κατόπιν. Έχουμε μια κοινή δήλωση των διαφόρων ΜΚΟ του πλαισίου επί του πλαισίου Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τη ΜΚΟ εδώ που συνεισέφεραν και στην έκθεση της Μάλιν αλλά και σε προηγούμενες εκθέσεις του πακέτου ασύλου και της έκθεσης για την επανεκατάσταση. Έχουμε λοιπόν την Πέτρα Χουκ, επικεφαλής της Διεθνούς Καθολικής Επιτροπής Μετανάστευσης να μας παρουσιάσει την άποψη των ΜΚΟ για την πρόταση της ε, Κομισιόν Πέτρα. Αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που η κυρία Μπιόκ και η Επιτροπή ΛΥΠΕ μας δίνει τη δυνατότητα να αφαιρθούμε στην πρόταση της Κομισιόν. Εμείς εργαζόμαστε με διάφορες ε, ΜΚΟ. Ε, πρόκειται για μια κοινή δήλωση Α, δεν νομίζω ότι 10 λεπτά αρκούν για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Οπότε θα τονίσω κάποια πράγματα. Να τονίσω ότι η ΜΚΟ που εργάζονται εδώ και καιρό στην επανεγκατάσταση και επιτόπου και στις χώρες ε, πρώτης ε, αναφήξεις και στα εθνικά προγράμματα για την υποδοχή και την ενσωμάτωση. Οι οργανώσεις λοιπόν είναι η Κάριτας Ευρώπα, η ΣΥΣΥΜΗ, e, η Επιτροπή των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μεταναστών και Εξορίστων, η Διεθνής Επιτροπή ε, Διάσωσης και το Ερυθρό Σταυρός και η δική μας οργάνωση βεβαίως. Έχουμε κοιτάξει διάφορα σημεία των προτάσεων. Και έχουμε κάποιες ανησυχίες, αλλά βεβαίως ε, τονίζουμε την ανάγκη του να υπάρχουν κάποια εναρμονισμένα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποιους ε, τομείς όπου μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Πρώτα απ' όλα, θα λέγαμε ότι το πλαίσιο δεν θα πρέπει να καταστήσει την επανεγκατάσταση υπό όρους, με όρο δηλαδή την συνεργασία των τρίτων χωρών. Θα πρέπει να δει τις ανάγκες ε, των καταστάσεων, της κατάστασης ε, διεθνούς προστασίας ε, και ατόμων τα οποία έχουν μείνει μερικές φορές και πάνω από 10 χρόνια σε στρατόπεδα προσφύγων παρατηρήσαμε ότι ο κανονισμός θα μπορούσε να είναι πιο διαφανός και θα πρέπει να δομηθεί πιο ξεκάθαρα. Και το βέβαια υπάρχει η παραδοσιακή επανεγκατάσταση υπό το πλαίσιο της ΥΠΑ του ΙΕ, αλλά και, και ένωση εσωτερικά εκτοπισμένων, οικογενειακή επανένωση, ανθρωπιστικές βίζες κτλ. Και βεβαίως μετά το να είναι κανείς ανάδοχος δεν είναι τρόπος τόσο επανεγκατάστασης, αλλά μάλλον χρηματοδότησης και εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή τα κριτήρια αυτά δεν είναι ευθυγραμμισμένα με το εγχειρίδιο της υπατσαρμοστίας του ΙΕ. Υπάρχει το πλαίσιο το οποίο θέτει δυσανάλογα και αφαίρετα κριτήρια για την επενεγκατάσταση προσφύγων και βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες προβλέψεις για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των προσφύγων. Για να επανέλθω σε κάποια από τα σημεία, το άρθρο 4 των σημείων που θα ληφθούν υπόψη ε, για να ληφθεί απόψη από πού θα γίνουν οι επανακαταστάσεις ε, σχετίζεται με στόχους διαχείρισης της μετανάστευσης, επανεισδοχή κλπ. Όπως ε, είπε και ο συνάδελφος από την Υπατή Αρμοστία του ΙΕ, η επανακατάσταση δεν είχε στόχο. Αυτό είναι ένα εργαλείο προστασίας και αλληλεγγύης και είναι αυτή η ερμηνεία σημαίνει μετακίνηση από τον ανθρωπιστικό στόχο που στόχο έχει να προστατεύσει ευπαθή άτομα και να τους δώσει μία μόνιμη λύση σε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε πως ε, οι καταστάσεις, οι μακροχρόνιες από ό,τι φαίνεται δεν περιλαμβάνονται εδώ πέρα. Η Κομισιόν μιλάει για τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι στην μεταναστευτική οδό προς την Ευρώπη. Δηλαδή τι κάνουμε με τους Κογκολέζους στην περιοχή των μεγάλων λιμνών της Αφρικής και άρα θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ανθρωπιστική ουσία της επαναγκατάστασης και να συνεχίσει να βασίζεται στις ανάγκες των πιο ευπαθών. Επιστρέφουμε τώρα στους στόχους του πλαισίου επανεγκατάστασης. Δεν αναφέρονται τόσο ξεκάθαρα. και βεβαίως ε, θα θέλαμε να υπάρξει αύξηση των βιώσιμων λύσεων, κάτι το οποίο βεβαίως περιέχεται στο πλαίσιο και κάτι το καλωσορίζουμε γιατί ξέρουμε άρα ποιες είναι οι φιλοδοξίε τη Ευρώπη, γιατί ο κανονισμός αυτός θα καθορίσει ένα πλαίσιο τα επόμενα 10-15 χρόνια οπότε πρέπει να υπάρχει ένα όραμα το οποίο δεν θα κοιτάει μόνο την τρέχουσα κατάσταση στην Τουρκία παραδείγματο χάρη αλλά θα έχει και μια πιο μακροπρόθεσμη άποψη άρα προτείνουμε το άρθρο 7 να περιλάβει στόχους αντί για αριθμούς και θα θέλαμε να γίνει ρητή αναφορά στις ε, ανάγκες που προβλέπει κάθε χρόνο η υπατερμοστία του ΙΕ και ένα ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια που είμαστε και μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσφύγων και Εξοδρίστων θεωρούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λαμβάνει ένα 25% των ατόμων που χρήζουν προστασία κάθε χρόνο παγκοσμίω. Αυτές θα μπορούσαν να είναι κάποιες πρώτες ε, φιλοδοξίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε For transparency reasons, we. I have a Swedish somewhere here. Okay. For transparency reasons, we would like. Για λόγους διαφάνειας. Ο κανονισμός καλύπτει και την παραδοσιακή, θα έλεγα, επανεγκατάσταση και άλλες νόμιμες διόδους όπως την ανθρωπιστική εισδοχή. Οπότε θα θέλαμε να εισαχθεί αυτό σε ολόκληρη την πρόταση και ειδικά τα άρθρα 2 και 8 να κάνουν αυτή την διάκριση για να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Κοιτώντας τώρα την επιλεξιμότητα για επανεγκατάσταση, βλέπουμε ότι το άρθρο 5 καθορίζει κατηγορίες προσφύγων που μπορούν να επανεγκατασταθούν με το προτινόμενο πλαίσιο, που δεν ανταποκρίνονται πλήρως με τις κατηγορίες της υπατσαρμοστίας του Παραδείγματος χάρη άτομα τα οποία δεν έχουν εναλλακτικέ διαρκείς λύσεις, δηλαδή δεν μπορούν να ενταχθούν τοπικά ή να επιστρέψουν στη χώρα τους, δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό. Άρα είναι ασαφές το εάν θα υπάρχει ε, επαναγκατάσταση για αυτά τα άτομα. Θα θέλαμε αυτό να αναφερθεί ρητός. Ο οργανισμός περιλαμβάνει άτομα με κοινωνικο-οικονομική ε, ευπάθεια, μια νέα κατηγορία που έχει επίσης εισαχθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ένας προς έναν με την Τουρκία και θεωρούμε πως θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη η πανεγκατάσταση με τα κριτήρια της ΥΠΑ στο του για την επανέναση οικογενειών που αναφέρθηκε ήδη από τον συνάδελφό μας θα θέλαμε να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε να διατηρηθεί αυτό το κριτήριο της περιπτώσεις όπου θα είναι η μοναδική περίπτωση βανούς οικογενειών. Το άρθρο 5 Β περιλαμβάνει άτομα τα οποία είναι ήδη παρόντα στην Ευρώπη και την δυνατότητα διατήρησης της οικογενειακής ενότητας. Αυτό δεν είναι οικογενειακή επανένωση. Και υπάρχει οδηγία του 2003 του Συμβουλίου για την Οικογενειακή Επανένωση. Τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας έχουν δικαίωμα στην ε, οικογενειακή επανένωση. Αυτός είναι άλλος ένας, ε, άλλη μια δίωδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δηλαδή η ίδια οικογενειακή επανένωση και το πλαίσιο της υπατσαρμοσίας του ΙΕ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλες περιπτώσεις. Άρα προτείνουμε να προσθεθεί στο τρέχον άρθρο 5β2 τέτοια άτομα μπορούν να ε, χρησιμοποιηθεί για τέτοια άτομα μόνο αν αυτό δεν είναι δυνατόν για μέσω άλλων ε, νομικών διατάξεων. Για την οικονομική στήριξη. Μόνο η επανεγκατάσταση που λαμβάνει η χώρα από περιοχές προτεραιότητας όπως αυτές αναφέρονται σε σχέδια προτεραιότητας ε, μπορεί να λάβουν στήριξη η οποία ανέρχεται σε 10.000 αν πρόσφυγα. Επίσης το ίδιο ισχύει και για την παραδοσιακή επανακατάσταση και για άλλους τρόπους, ε, τύπους εισδοχής. Αυτό ίσως αποθαρρύνει τα κρατημέλη από το να συνεχίσουν ε, τα υφιστάμενα προγράμματα επανακατάστασης που θεωρούμε ότι είναι η βάση της ε, παράδοσης της επανεγκατάστασης στην Ευρώπη. Επίσης η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ευέλικτη για να επιτρέψει στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό προσφύγων να μετακατασταθούν εξαρτήτως του εάν είναι σε περιοχή προτεραιότητας και αυτό θα ισχύσει ιδιαίτερα θα πρέπει να ισχύσει ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη επίγουσας προστασίας και επίγουσας επανεγκατάστασης. Οπότε θα πρέπει να έχουμε αυτή την διτή προσέγγιση που υπάρχει στο τωρινό ε, ΑΜΙΦ, το Ταμείο Σύλλου Μετανάστευσης και Ένταξη, όπου τα κράτη-μέλη λαμβάνουν 10.000 ανά άτομο και 6.000 για άτομο εκτός των προτεραιοτήτων. Έτσι γινόταν στο παρελθόν. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει, αλλά θεωρούμε ότι οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να διατηρήσουν το ότι ε, θα έχουμε ως δυνατόν περισσότερους που θα γίνονται δεκτοί. Και βέβαια θα μπορούσαν να λαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις ε, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η επανεγκατάσταση έτσι θα σώζει ζωές και αυτή είναι νομίζω μια μεγάλη συνεισφορά παγκόσμια της ευρωπαϊκής επανεγκατάστασης. Αναφέραμε ήδη τις δυσανάλογες κατηγορίες που αποκλείονται, που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στον κανονισμό. Άτομα τα οποία έχει αρνηθεί ένα άλλο κράτος μέλος να επανεγκαταστήσει Και βεβαίω αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε διαδικασία επιλογή από κράτη σημαίνει ότι κάποια άτομα επιλέγονται και κάποια δεν επιλέγονται. Δηλαδή απορρίπτονται περιπτώσεις για διάφορου λόγου. Μπορεί παραδείγματο χάρη κάποιο να έχει, ιατρι... Ε, έχει μια ασθένεια για κατά το οποίο σημαίνει κόστο που δεν θα θέλει να καλύψει ένα κράτο. ή να μην διαθέσει στέγαση για μια μεγάλη οικογένεια αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούν μετά να αποκλειστούν στο μέλλον από άλλες χώρες από το να επανεγκατασταθούν. επειδή απλά απορρίφθηκαν μια φορά στο παρελθόν. Επίσης, όπως είπαν και οι συναλφοί μας από την Υπατήρμοστία του ΟΗΕ, το πλαίσιο θα πρέπει να βασιστεί στις υφιστάμενε διαδικασίες. Τα άρθρα 10 και 11 περιγράφουν τι διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν και έτσι θα αναθεωρηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο που ορίζει στο άρθρο 10 ότι η καταγραφή και ταυτοποίηση θα γίνεται από κράτη-μέλη αντί για την υπαδιαρμοστία του ΟΗΕ. Τα κράτη-μέλη θα γίνουν αυτοί οι οποίοι κυρίως θα διαχειρίζονται όλες τις στοιχείες των προγραμμάτων εισδοχής οι διάφορες πτυχές ε, που αφορούν στην ε, ταυτοποίηση αυτή τη στιγμή είναι ασαφείς αντί να, εστιάζουν στην εισδοχή τα κράτη-μέλη τώρα θα εστιάζουν στην ταυτοποίηση και την επεξεργασία των αιτήσεων και βεβαίως η πρόταση από ό,τι τυποποιεί κάποιες διαδικασίες που είχαν αναπτυχθεί στην ε, συμφωνία με την Τουρκία ναι, τελειώνω. Όσον αφορά τις επιταχυμένες διαδικασίες, νομίζω αναφέρθηκε η κατεπίγουσα επαναγκατάσταση, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα ήθελα απλά να πω σύντομα για το θέμα της υποδοχής και της ένταξης. Εάν ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο σύστημα υποδοχής σε ολόκληρη την όναση, ο κανονισμός θα πρέπει να δει ένα σχεδιασμό προαναχώρησης ήδη. Οι διαφορές θα υπάρχουν πάντα μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την στήριξη και τις οικονομικές ευκαιρίες, όμως πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί έτσι ώστε να υπάρχει ε, έτοιμη υποδοχή στις χώρες που θα, δεχτεί, θα δεχτούν τις προσφύγες. Θα υπάρξει δηλαδή και μια πρώτη ενημέρωση. Επιπλέον τιμωρούνται όσοι πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη, αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες. Ο κανονισμός άρα δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα για το οποίο συχνά δεν πετυχαίνει η επαναγκατάσταση. Όσον αφορά την ένταξη, οι προσπάθειες αυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ζητάμε άρα τα κράτη-μέλη να απαιτείται να προγραμματίζουν τα κατάλληλα προγράμματα για την υποδοχή των προσφύγων. Αυτό πρέπει να γίνει σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές στο τοπικό επίπεδο και με επαρκή χρηματοδότηση. Η επαναγκατάσταση είναι μια εταιρική δραστηριότητα που απαιτεί συνεργασία από τον ΟΗΕ, τα κράτη-μέλη και την κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών βρίσκεται εδώ για να συνεργαστεί πλήρως για να γίνει ε, επιτυχής η επαναγκατάσταση στην Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω αυτά Περνάμε κατευθείαν στον κύριο Όσκαρ Εκπλατ από το Σουηδικό Οργανισμό Μετανάστευσης που θα μας παρουσιάσει το Σουηδικό, το εθνικό πρόγραμμα δηλαδή επανεγκατάστασης. Έχετε το λόγο για 10 με 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας που με κάλεσε για να μιλήσω για κάτι διαφορετικό, όχι για την πρόταση του κανονισμού, γιατί προσωπώ μια, έναν οργανισμό μετανάστευσης και θα σας παρουσιάσω την εμπειρία του Εθνικού Οργανισμού μετά από 70 χρόνια του προγράμματος επανεγκατάστασης που εφαρμόζουμε στη Σουηδία. Θα εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε αρκετά επιτυχείς παρόλο που γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εφαρμόσει κανεί την επανεγκατάσταση. Και σίγουρα και αυτή η πολυμορφία στις μεθόδους ε, δεν είναι κακή. Θα ήθελα να δηλώσω αυτής εξ αρχής ότι η επανεγκατάσταση είναι ε, κάτι που προϋποθέτει μεγάλο φόρτο εργασίας. Όχι τόσο ένταση πόρων, αλλά τεράστιες προσπάθειες συντονισμού και πλούσια πείρα για να είναι αποτελεσματική. Έχουμε δέκα ουσιαστικά ε, συνομιλητές φορείς, ώστε να φτάσει κάποιος ε, από τη χώρα του στη Σουηδία και μέσω του συντονισμού και των, της Έχω ήδη πλούσια πείρα από να ασχολήσει με το θέμα αυτό και ελπίζω να συνεχίσω να ασχολούμαι για άλλα τόσα χρόνια, άλλα 13. Τώρα, το σουηδικό πρόγραμμα ε, προβλέπει 1.900 θέσεις και για το χρόνο προβλέπουμε 3.400 για το 2017 και για το 2018 η κυβέρνηση προβλέπει 5.000 πρόσφυγες που θα υποφελούνται από αυτό το πρόγραμμα. Σημαντική αύξηση δηλαδή. 163.000 ήταν οι αιτούντες άσυλο πέρυσι μόνο. Βέβαια, ε, αυτό γίνεται στα πλαίσια των αναγκών ε, και της αυτοποίησης που κάνει η πατερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση με την ε, νομολογία, με τις πολιτικές, με τα Ένωμα συστήματα προστασίας και παροχής ασύλου της Σουηδίας και μετά την ε, θέσπιση νέων κανόνων το καλοκαίρι προβλέπεται εξαίρεση από, το, από τη διάρκεια παραμονής ε, που είναι μόνιμη για τους επανεγκαταστημένους. Εδώ παρουσιάζω τις αδερές γραμμές ε, του προγράμματός μας. Χαιρόμαστε που υπάρχει. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε διάφορε προκλήσει. Θα ασχοληθώ με αυτέ αργότερα. Στηρίζουμε το πρόγραμμά μα ε, στην αξιοπιστία και στη συνοχή και την ε, συνέπεια. Ε, το πρόγραμμά μα ισχύει από το 1950, από τη δεκαετία του 50. Έχει γίνει γενικώ αποδεκτό από το κοινό στη Σουηδία και είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο και για την υπατερμοστία αλλά είναι αξιόπιστο εργαλείο και για τους ε, δήμους, για τις περιφερειακές αρχές, γιατί τέτοιου είδους ε, ε, επιχειρηματικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις περιφέρειες για να αναπτύξουν και τη δική τους εμπειρογνωσία. Επίσης και για μεμονωμένους πρόσφυγες είναι συνεπές και αξιόπιστο γιατί παρέχει μόνιμη προστασία. Ε, ο οργανισμός μας λαμβάνει εντολή από την κυβέρνηση και στηρίζουμε το έργο μας σχεδόν αποτελεσματικά στην αξιολόγηση αναγκών της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Και κάθε χρόνο αποφασίζουμε για την κατανομή των σουηδικών ποσοστώσεων, αλλά με βάση το έγγραφο για τις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης που ε, κάθε καλοκαίρι δημοσιεύει η αρμοστία του ΟΗΕ. Και μάλιστα τώρα ετοιμάζονται ε, τα έγγραφα για το νέο γύρο επανεγκατάσταση. Οπότε η αξιολόγηση των αναγκών που κάνει η πατερμοστία έχει θεμελιώδη ρόλο στι δικέ μα ποσοστώσει και μάλιστα αφορά και τι υπεμονωμένε περιπτώσει. Γιατί στηρίζουμε όλο μα το έργο στην αδυναμία του δικού μα οργανισμού να αποφασίζει μεμονωμένα για το ποιο πρόσφυγα θα πρέπει να υποβληθεί στο σουηδικό πρόγραμμα επανεγκατάσταση και ποιο εκπίπτει. Και μάλιστα αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του οργανισμού μας, γιατί έτσι μας ε, ε, απαλλάσσει από συζητήσει ε, με μεμονωμένους, με συγγενείς για το ποιος είναι δικαιούχος τέτοιου δικαιώματος επανεγκατάστασης. Αυτό το ρόλο τον αναθέτουμε στο, στην ύπατη αρμοστία. Το σχετικό πρόγραμμα είναι πολύ μορφό από γεωγραφική άποψη και καλύπτει όλες τις υπήρους. Βέβαια, κυρίως επικεντρώνεται τώρα στη Συρία. 40 με 50% των δικαιούχων επανεκατάστασης του Σουηδικού Προγράμματος επανεκατάστασης είναι Σύριοι. Χρησιμοποιείται όμως το πρόγραμμά μας και για άλλες περιπτώσεις, ε, για τους Αφγανούς στο Ιράν, για τους ε, Κενιάτες, για τους Ερυθρέους ε, στο Σουδάν, ένα θέμα που δυστυχώς δεν συγκεντρώνει μεγάλη προσοχή παγκοσμίω. Οπότε ασχολούμαστε και με έκτακτες ε, καταστάσεις, αλλά και με παραταμένες ε, καταστάσεις για πρόσφυγες που για μεγάλο χρόνο βρίσκονται σε καθεστώς χωρίς να έχουν λάβει το δικαίωμα επανεγκατάστασης. Επίσης, έχουμε τη μεγαλύτερη υποποσόστοση για έκτακτες περιπτώσεις στον κόσμο. Φέτος ε, οι 50, του χρόνου θα είναι περισσότεροι και παρέχουμε και ε, ειδική προστασία σε όλους, σε εκείνου είτε αντίρρησης αντιφρονούντες ή ως φοβούνται επικείμενη δίωξη ή που έχουν κάποια σοβαρή νόσο που τρέχουν κίνδυνο να πεθάνουν ή να υποκύψουν στις αρνητικές συνέπειες της νόσου τους αν δεν επανεκατασταθούν όταν αντιμετωπίζουν άμεση επαναπρόθεση στη χώρα τους ε, στην οποία απειλούνται με βασανιστήρια θανατική ποινή και βλέπουμε ανθρώπους ε, που πραγματικά μπορούμε να τους βοηθήσουμε από αυτή την άποψη. Βέβαια, όχι πάντα, γιατί πολλές φορές ο χρόνος ε, είναι αντίπαλός μας και βλέπουμε εδώ την αρνητική πλευρά και δυστυχώς δεν μπορούμε να σώσουμε όλους όσους θα θέλαμε. Το σύστημά μας ε, ε, εφαρμόζεται διακρίτως ε, με βάση τους κανόνες της οδηγίας αναγνώρισης και τον, τη συνθήκη του ΟΗΕ για την επικουρική προστασία. Δύο είναι βασικοί παράγοντες για την επιλογή κάποιου για το σουηδικό πρόγραμμα. Δεν έχουμε ειδικέ ομάδες, πέραν τη γεωγραφική κατανομή που ζητάει η πατιαρμοστία. Δεν έχουμε ε, ιδιαίτερη εστίαση σε, σε φύλλο, σε ηλικιακέ ομάδες, σε εθνότητα ή σε θρησκεία. Επίσης το πρόγραμμά μας ε, είναι πολύ ελαστικό, ευέλικτο και έχουμε στενή συνεργασία με την υπετερμοστία ώστε να προσαρμοζόμαστε στις ε, ε, ανάγκες που μεταβάλλονται συνεχώς. Βέβαια, ως ε, κυβερνητικός ε, υπάλληλος χρησιμοποιούμε τη δημοσιονομική χρήση, αλλά μέσα σε αυτή τη δημοσιονομική χρήση πολλά αλλάζουν. Και ακριβώς θέλω αυτή την ελαστικότητα για να μπορούμε να αλλάζουμε την εστίασή μας. Το 2011 είχαμε τη Λιβύα, τώρα έχουμε Συρία και τους εσωτερικά εκτοπιστέντες εντός της Συρίας που χρήζουν προστασίας, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και άλλες χώρες. Η ελαστικότητά μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευελιξία και των Δήμων και Περιφερειών που υποδέχονται και άλλους από αυτούς που αρχικά είχαν προγραμματιστεί να υποδεχθούν. Έτσι έχουμε περιπτωσιολογική ανάλυση με, σε συνεργασία με τους Δήμους. Επίσης έχουμε μια καλά εφοδιασμένη υπηρεσία που πολύ με πολύ ταχείες διαδικασίες εξετάζει τις ε, περιπτώσεις, σταματά υποθέσεις που δεν έχουν μέλλον, αλλά και ε, διεκπερώνει γρήγορα υποθέσεις που φέρουν τα κριτήρια για να προχωρήσουν. Προϋπολογισμός, κάτι που ενδιαφέρει πολλούς συνήθως. Η επανεκατάσταση θεωρείται για πολλούς ότι απορροφά πολλούς πόρους. Βλέπετε το ανοιχτό γαλάζιο τμήμα του κύκλου, που είναι το κόστος για μία διετία στη Σουηδία, που είναι ακριβώς το ίδιο επίδομα που δίνεται στους Δήμους για όσους φτάνουν στα πλαίσια του καθεστώτος ασύλου. Το σκούρο μπλε είναι το επιπλέον κόστος της επανεγκατάστασης, η ανάγκη σε προσωπικό και οι επιμελητιακές ανάγκες. Για μετάβαση αποστολών, για την ε, ε, μεταφορά των ε, προσφύγων στη Σουηδία και το καθεξής. Προκλήσεις. Στέγασε φυσικά η μείζον πρόκληση, όχι μόνο στη Σουηδία, παντού. Ε, το χρόνο θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό και η παροχή στέγης για τους νέους ε, πρόσφυγες είναι μεγάλη πρόκληση. Θέλουμε να βρούμε καινοτόμους τρόπους και ευρηματικούς, ώστε στη συνεργασία με τους Δήμους να βρούμε τρόπους να στεγάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, ε, άδειες, ε, επιμελητιακά ζητήματα, πώς θα φέρουμε, μεταφέρουμε ανθρώπους από την άλλη άκρη του φορές. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και το, εθνικό δίκτυο, το παγκόσμιο δίκτυο ε, μετανάστευσης είναι σημαντικός εταίρος. Ε, πολιτισμικός προσανατολισμός. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα πρέπει να ξέρουν ε, οι πρόσφυγες σε τι κοινωνία θα ενταχθούν, τι να περιμένουν από το ταξίδι τους, από τον καταβλισμό των προσφύγων στην νέα κοινωνία. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα της ενημέρωσης θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο διεξοδικά και είναι το ίδιο του συστήματος, αλλά από πιο σημαντικά. Γι' αυτό θα πρέπει να το αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Το θέμα της ασφάλειας και του αποκλεισμού, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μεριμνούμε γι' αυτό και στα θέματα της επανεγκατάστασης. Και έχουμε παρόμοια ανάλυση με τις υπηρεσίες ασφάλειας για την επανεγκατάσταση. Και φυσικά είπα ότι η αρμοστία κάνει μια πολύ καλή προεργασία και αποτρέπει μερικές, μερικούς κινδύνους και απειλές για την εθνική ασφάλεια. Οπότε γενικώ η επανεγκατάσταση είναι ασφαλής. Τέλος, η Σουηδία ίσως δεν είναι η καλύτερη χώρα παράδειγμα για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, γιατί υπάρχει ισχυρό κρατικό μονοπόλιο για την παροχή υπηρεσιών. Έχουμε να διδαχθούμε από άλλε χώρε περισσότερο τη Ευρώπη για την ανάπτυξη νέων ιδεών, για συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και συνεργασία με Δήμου και περιφέρειε. σω εκεί δεν είμαστε το παράδειγμα προ μίμηση ό,τι αφορά τη συνεργασία κράτου και περιφερειακών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ίσως όμως ε, θα μπορούσαμε με διεθνή συνεργασία να αναπτύξουμε το δυναμικό της κάθε χώρας και έχουμε και ένα ε, σχέδιο ευρωπαϊκό ώστε να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα, ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να αντιμετωπίσει καλύτερα την επανεγκατάσταση. Επίσης, Έχουμε και εδώ καιρό μηχανισμό στήριξη σε σχέση με το ΑΕΡΑΜ και το Ηνωμένα Έθνη για να στηρίξουμε νέε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν χώρε επανεγκατάσταση και αφιερώνουμε κονδύλια στο θέμα αυτό αλλά και ε, παροχή εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστούμε πολύ που μας εξηγήσατε τι ακριβώ συμβαίνει στη Σουηδία. Περνάμε αμέσω τώρα στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση για να μας πει και την αξιολόγησή του για το προτινόμενο ε, πλαίσιο. Ένα τεταρτάκι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και λίγο, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουν οι συνάδελφοι να θέσουν τις ερωτήσει τους. Αν μπορεί ο συνάδελφο λοιπόν να μιλήσει σε 10 λεπτά μόνο. Πατρίς Κεσάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή πολλά σημεία τα έφυξαν ε, ήδη οι προλαλήσαντες, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω κάποια εξ αυτών. Είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Η δημιουργία ενός ε, πλαισίου ε, επανεγκατάστασης είναι κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και χρόνια πέραν της υποστήριξης προς τα εθνικά προγράμματα με τους εταίρους που βρίσκονται εδώ. Ξέρουμε ποιο πλαίσιο οδήγησε κατεπηγόντως να ε, δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα πλαίσιο για να ε, διασφαλίσει την προστασία και να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια στις πιο ευπαθείς ομάδες. Ε, και θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πρόσδεκτη η δυνατότητα να σχολιάσουμε το σχέδιο του πλαισίου, αλλά όπως και ο συνάδελφος από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία θα θέλαμε να επισημάνουμε και κάποια σημεία που θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ε, δώσει ένα σχέδιο συστάσεων προς την εισηγήτρια και σε εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τα χαράς να τα μοιραστούμε και μαζί σας. Όσον αφορά τους όρους, γιατί θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί πρόεδρος ε, σε πολύ σημαντικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τους κανόνες υποδοχής, τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνται και το καθεστώς ε, το οποίο θα ε, δίνεται στους πρόσφυγες αματιαθήξη τους. Επίσης, ε, οι γεωγραφικές προτεραιότητες βάσει συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και ασύλου αυτό θα μπορούσε ίσως να υποσκάψει τις αρχές που διέπουν ένα από τα πιο σημαντικά ανθρωπιστικά μέσα για να παρέχουμε ε, διεθνή προστασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενθυμίσουμε ότι η επανεγκατάσταση είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές μόνο για ένα κλάσμα των εκτοπισμένων ανθρώπων και των ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται από διάφορες ε, ε, διαδικασίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διάρθρωση μεταξύ του πλαισίου επανεγκατάστασης ε, και ε, των υφιστάμενων προγραμμάτων θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να μην είναι το ένα εις βάρος του άλλου. Ε, για να το πω διαφορετικά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο αριθμό των θέσεων που προσφέρονται θα είναι αξιόπιστος και ουσιαστικό, ιδίω αν είναι μια ασφαλή και νόμιμη εναλλακτική λύση σε άλλε διαδικασίε. Αυτή τη στιγμή από το σχέδιο πρόταση δεν φαίνεται να υπάρχει ένα ελάχιστο αριθμό στόχο, αναφέρεται απλώ ε, η βαθμιδόν κλιμάκωση των προσπαθειών, δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώ θα είναι αυτό, αλλά χωρί να επενδύξουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που θα επανεγκαθίσταται, δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό. Όσον αφορά τις αιτήσιες ποσοστώσεις για τα άτομα που επανεγκαθίσταται, ε, θα είναι αβέβαιο εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποσόστοση και φυσικά αυτό επηρεάζει και το έργο των άλλων εταίρων επιτόπου κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Ένα τρίτο σημείο το οποίο θα θέλαμε να θίξουμε όσον αφορά τις δευτερογενείς μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι πιστεύουμε ότι η σύγκληση μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων επαναγκατάστασης και η κοινή προσέγγιση είναι αυτά τα οποία θα βοηθήσουν να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τις δευτερογενείς μετακινήσεις, αλλά θα μπορέσει να έχει αποτέλεσμα μόνο εάν ευθυγραμμίσουμε συγγνώμη, τα δικαιώματα αυτών που έρχονται ε, και αυτών που την χάνουν διεθνού προστασία, και αυτό ε, με βάση και τον ε, αναθεωρημένο κανονισμό για τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό λοιπόν θα βοηθήσει και τα θέματα της μετανάστευσης και τις διάφορες πρακτικές και δεύτερον, Πέραν του γεγονότος ότι θα πρέπει όλοι να την χάνουν αντίστοιχο καθεστώτος, ε, τα άτομα τα οποία την χάνουν επανεγκατάσταση θα πρέπει να έχουν και αντίστοιχε διαδικασίες υποδοχής και προγράμματα ένταξης. Και εδώ έρχομαι στο τέταρτο σχόλιο μου για την ένταξη τρόπον την να, η ένταξη είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει να μην υπάρχουν πάρα πολλές ε, μετακινήσεις ε, δευτερογενώς, αλλά ε, η ένταξη είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει, είναι ο βασικός στόχος στο ανθρωπιστικό ε, πρόγραμμα και είναι και το κριτήριο για να μετρήσουμε την επιτυχία του προγράμματος. Θα θέλαμε λοιπόν να προτρέψουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτό το ε, πλαίσιο επανεγκατάστασης για να επικεντρωθούν περισσότερο στην ένταξη των ατόμων αυτών, όπως τόνισε και ο συνάδελφος από τη Σουηδία πρόκειται για μια ε, δαπανηρή διαδικασία που απαιτεί και συγκεκριμένε επενδύσεις υπάρχει ένα καταποκοπή ποσό 10.000 ευρώ. Ε, θα πρέπει εδώ να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι απλώς ένα κίνητρο. Μπορεί να καλύψει ε, το αρχικό κόστος, ε, αλλά δεν μπορεί να καλύψει την ένταξη, διότι χρειάζεται μακροπρόθεσμη δέσμευση και συγκεκριμένε δομές για να το επιτύχουμε. Η Σουηδία επίσης ε, είπε ότι ορισμένες φορές ε, παρέχουμε δυνατότητες επανεγκατόστασης και ένταξη ε, οικογένειες οι οποίες είναι τραυματισμένες και έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και παρά το γεγονός ε, ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έχουμε μέτρα πρώτης αναχώρησης, ε, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το να ε, καθορίσουμε τη διάρκεια ε, παραμονής προτείνεται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο τριών ημερών για να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα, να τους εξηγήσουμε και να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε και τις συνέπειες των επιλογών κάποιων να υπαναχωρήσουν την τελευταία στιγμή. Πρέπει επίσης να γίνονται κάποιες αξιολογήσεις αλλά ε, το να ε, μην υπάρχουν ε, μέτρα πριν ε, την αναχώρηση σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι επιτόπου. Ε, οι συνάδελφοι έκαναν και άλλα σχόλια. Ένα μεγάλο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων που έχουν φύγει από τη χώρα του χρειάζονται και αυτή η διεθνή προστασία και βρίσκονται εντό τη ίδια χώρα. Επομένω θα πρέπει να το δούμε και αυτό στο σχέδιο τη πρόταση. Για παράδειγμα, χώρε όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδά κάνουν εσωτερική επανεγκατάσταση στο παρελθόν ε, και την κάνουν εδώ και αρκετά χρόνια, Επομένω, δεν πρόκειται για κάτι καινοφανέ. Όσον αφορά το πλαίσιο, το πλαίσιο για να βρίσκουμε εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα για επανεγκατάσταση θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλο και χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας για να προλάβουμε περιπτώσεις διακρίσεων. Και επίσης δεν ξέρουμε κατά πόσο η επανεγκατάσταση είναι πάντα η κατάλληλη λύση για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Πιστεύουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση εάν υπάρχουν δυνατότητες ε, επανεγκατάστασης για εσωτερικά εκτοπισμένους, θα πρέπει να δούμε ε, κατά προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα άτομα και θα πρέπει όλα να γίνονται και βάση τη αιτήσει αξιολόγηση για τι ανάγκε, τη ΥΠΑ τη αρμοστία για τους πρόσφυγε. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλοξιμότητας και για να μην υπάρχουν διακρίσει και πάλι, ε, το οποίο δεν συνάδει και με ένα ανθρωπιστικά πρόγραμμα, ε, το οποίο θα πρέπει να διέπεται από ανθρωπιστικές αρχές, θα πρέπει ε, να συστήσουμε να μην υπάρχει το κριτήριο του αποκλεισμού, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε, ε, δεν δίνεται πρόσβαση ασύλου σε άτομα τα οποία αποπειράθηκαν αρκετέ φορέ να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποκλείσουμε και άτομα τα οποία είναι πολύ ευάλωτα, ε, επειδή απλώς και μόνον ε, επιχείρησαν να εισέλθουν ε, παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα προγράμματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έχετε προσκαλέσει και άλλες διεθνείς οργανώσεις στην ε, Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Επανεγκατάσταση και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους εγκαίρως, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς τη συζήτηση ε, με τη μακρά πείρα που έχουμε στον τομέα αυτό και φέτος άλλωστε έχουμε και τα 65 χρόνια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης σε θέματα αυτά. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι ο μηχανισμός ε, τριμερού συντονισμού της ΥΠΑ Αρμοστίας ε, μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της ΥΠΑ Αρμοστίας θα πρέπει να γίνεται σεβαστός και να ενισχύσουμε και το ρόλο του, διότι ελοχεύει ο κίνδυνος αν δημιουργήσουμε μια ε, παράλληλη δομή να μην είναι αποτελεσματική. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να σχολιάσουμε. Θεωρούμε ότι είναι πολύ ε, καλοδεχούμενη αυτή η πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επανεγκατάστασης και θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κεσάντα και ευχαριστώ που ήσταν σχετικά σύντομος. Περνάμε στη συζήτηση τώρα. Ε, η κυρία Μάλιν Μπιόρκη, συγγήτρια, θα αντιλήσει κάποια συμπεράσματα μετά το πέρας ζήτηση. Όποιοι θέλουν το λόγο, στο δηλώσουν. Βλέπω κάποιους και οδησηγητές και δύο μέλη της Επιτροπής που έχουν ζητήσει το λόγο. Άλλος κανείς. So, um, Ξεκινάμε με την κυρία Stevens. Eh, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Σας ευχαριστώ για την εμπειρία που μας μεταφέρατε και τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις σας. Έχω δύο ερωτήσεις ε, για, εσά, για την υπατήρμοστια του Ιέλα να σας πω. επειδή σε αρχής σύμφωνη με την πρόταση. Η πρόταση έχει στόχο να συνδέσει όλες αυτές τις εθνικές προτάσεις και να δημιουργηθεί μια θέση διαπραγματευτική σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα συγκεντρώσει τις εθνικές ανθρωπιστικές της ε, προσπάθειες, αλλά ε, στο στυλ της συμφωνίας με την Τουρκία και έτσι θα υπάρξουν θέσεις οι οποίες θα προβλεφθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και επιδοτήσεις για κέντρα υποδοχής. Θα ήθελα να θέσω τώρα δύο ερωτήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι η πατερμοσία του ΙΕ έχει ένα σύστημα point system ε, για να κρίνει ποιοι είναι οι πιο ευπαθείς ε, πρόσφυγες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το πλαίσιο προσθέτει δύο νέες κατηγορίες, δηλαδή οικονομικούς ε, μετανάστες και την επανένωση της οικογένειας. Τι άποψη έχετε για αυτές τις προσθήκες και ποια θα είναι η πρακτική, ο πρακτικός αντίκτυπος στην καθημερινή κατάσταση. Σας ευχαριστώ. τι πέρι. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα κάποιον να λέει ότι η σύνδεση της πρότασης επανεγκατάστασης όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για, με τη συνεργασία με τρίτες χώρες είναι καλή ιδέα, εκτός αν μου ξέφυγε. Αλλά νομίζω πως είναι κάτι το επικίνδυνο αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που μετεγκαθίστανται στην Ένωση. Θα με ενδιαφέρει να το ακούσω να ακούσουμε τη θετική πτυχή. Όσον αφορά την χρηματοδότηση και ανέφερε κάτι η τελευταία μιλήτρια, έχετε κάποια εμπειρία ε, ότι δηλαδή η χρηματοδότηση θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο, ενώ ξέρουμε ότι το κόστος για αυτούς τους ανθρώπους θα είναι πολύ περισσότερο από τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο λειτουργεί αυτό κατά την άποψή σας μετά. Ε, μία ερώτηση στον ε, κύριο από τη Σουηδία. Εξηγήσατε ότι χρειάζεται πολλή ε, δουλειά, είναι μια υπόθεση έντασης εργασίας η επαναγκατάσταση. Εμείς λοιπόν οι προοδευτικοί στο Κοινοβούλιο σκεφτόμαστε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή 250.000 άτομα το χρόνο με την εμπειρία σας λοιπόν που εσείς ε, εγκαταστάτε άτομα τόσο καιρό. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να καταφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ή εμείς οι προοδευτικοί είμαστε κάπως φιλόδοξοι. Ελπίζω όχι, ελπίζω να μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τέλος, είναι σαφές οπωσδήποτε, πως είπατε, η το παίζει ένα ρόλο κλειδί σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά υπάρχουν κάποια μέρη, η Τουρκία παραδείγματος χάρη, όπου η πατεραμοστία του ΟΗΕ δεν είναι ο οργανισμός ο οποίος καταγράφει τους Σύριους παρά μόνο τους Ιρακινούς και λοιπούς που είναι πολύ λιγότεροι. Η πατερμοστία του ΟΗΕ λοιπόν απαιτείται πάντα να είναι ο συνομιλητής όταν μιλάμε για επαναγκατάσταση ή θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γνωρίζοντας βεβαίως πάντα την αξιολόγηση των αναγκών που υπάρχουν. Και είναι παγκόσμιες προδιαγραφέ. Ευχαριστώ, Κέιτ. Ως απάντηση προς την ερώτηση των βουλευτών. Είπαν και κάποιοι συνελφοί ότι ήθελαν επίσης να απαντήσουν. Λοιπόν, Σαρτζεντίνη κατόπιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ανησυχώ για την πρόταση αυτή και δεν είμαι σίγουρη για το εάν θα οδηγήσει σε επανεγκατάσταση περισσότερων ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα το πάνελ να μου εξηγήσει τις σκέψεις του. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξουν νόμιμες διόδη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να αυξηθεί ουσιαστικά και άκουσα κάποιον που είπε ότι πρέπει να πάρουμε 25% των ατόμων ε, παγκοσμίω κατέτος, Θεωρείτε πως η πρόταση αυτή επιτάπητος οδηγεί σε αύξηση των αριθμών. Θεωρείτε πως βλέπετε την εναρμόνιση των προδιαγραφών μας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς το βλέπετε αυτό υπό το φως των εθνικών πολιτικών που υπάρχουν. Μία από αυτές τις πτυχές ε, που με ανησυχεί είναι η πρόταση ότι μπορεί να απορριφθεί κάποιος και δεν χρειάζεται να πούμε στα άλλα κράτη-μέλη ποιος ήταν ο λόγος της απόρριψης και το σκεπτικό είναι ότι οι υπόλοιποι 27 δεν μπορούν ούτως ή άλλως να τον να εγκαταστήσουν. Ίσως η πατερμοστή του θα μπορούσε να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει με αυτές τις περιπτώσεις ή να βρει κάπου αλλού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είπα αυτό το φως. Πώς ε, βλέπετε την νομοθεσία που προτείνεται Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ. Κυρία Βινμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες. Νομίζω ότι όπως θα είδατε, εμείς στη Σουηδία έχουμε εφαρμόσει την επανεγκατάσταση με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και νομίζω ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την ύπατη αρμοστία και να βοηθήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν από τον κίνδυνο και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σκέφτηκα και κάποια πράγματα. Πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει το πλαίσιο Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε επανεγκατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα θα υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού πλαισίου, του πλαισίου που υπάρχει σε εθνικό πλαίσιο. Επομένως, ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των δύο. 10.000 ευρώ για κάθε επανεγκατάσταση, για κάθε άτομο το οποίο επανεγκαθίσταται, θα καταφέρουμε να έχουμε επανεκατάσταση περισσότερων ατόμων. Ναι, μεν, αλλά σκέφτομαι και τις συνέπειες ε, όσον αφορά τη, ο προσωπικό, ε, τι πόρους χρειαζόμαστε για να εφαρμοστεί ε, το πλαίσιο πέραν του οικονομικού. Ε, όσον αφορά τα κριτήρια, αναφερθήκατε σε διάφορα κριτήρια, γυναίκες εγγύους, ε, γυναίκες με παιδιά, ε, βασανισμένα άτομα κλπ. Αλλά υπάρχει ένα κριτήριο που λέει ότι μπορεί να είναι άτομα το οποίο μπορεί να είναι ευάλωτο κοινωνικο-οικονομικά. Τι θα πει αυτό το κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτο άτομο. Στην πλειοψηφία τους τα άτομα τα οποία ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων είναι κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτα. Ε, πώς θα κάνουμε τη διάκριση. Επίσης, θεωρείτε ότι ε, θα υπάρχει επανακατάσταση από την Ιταλία και την Ελλάδα προς άλλα κράτη-μέλη, ας πούμε, σε πρώτη φάση. Ε, τι άποψη έχετε για τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ε, λαμβάνετε υπόψη σας και την κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σκεφτόμουν ότι ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μας κάνει κάποια σχόλια. Καταρχήν θέλει άλλος κανείς το λόγο από τα μέλη της Επιτροπής. Όχι. Οπότε, από την IRRC. Και ανέφερα την IRC γιατί αναφερθήκατε στο πρόγραμμα και είπατε ότι θέλετε το λόγο και το ίδιο έκανε και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και κυρίως την Πέτρα και την ICMC για την τεράστια προσπάθεια που έκανε για να συγκροτήσει αυτή την κοινή διακήρυξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η παρέ, παρά, παρέχει έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια ε, και έχουμε και εκτεταμένες ε, επιχειρήσεις ε, και εμπειρογνωσία, πολιτική, εμπειρογνωσία σε πολιτική επανεγκατάστασης και βοηθούμε χώρες στα προγράμματά τους επενεγκατάστασης. Εδώ και καιρό ζητούσαμε ένα παρευρωπαϊκό σύστημα και πρόγραμμα επενεγκατάστασης γιατί είναι μια πλούσια περιοχή και ανθρωπιστικό παράγοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταπεξέλθει στι διεθνεί υποχρεώσει τη. Και όπω και άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, θέλουμε να είναι αξιόλογο το σύστημα και να μην υπόκειται σε περιορισμού. Θα πρέπει να είναι επίση ένα συμπληρωματικό εργαλείο που δεν θα εκτοπίζει άλλε αυθόρμητε αφήξει ή άλλε άλλες όπως είπε και η Πέτρα, είναι σημαντικό το πλαίσιο επανεγκατάστασης να οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των προσφύγων που επανεγκαθίστανται στην Ευρώπη και να μην ε, θεσπίσει ανώτατα όρια επανεγκατάστασης. Επίσης, η Άρση ζήτησε τουλάχιστον 540.000 ε, ε, πρόσφυγες να επανεγκατασταθούν στην επόμενη πενταετία, 108.000 ε, δηλαδή ε, πρόσφυγες στον χρόνο. Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και εφικτό κάτι τέτοιο και στα, στις διάφορες μελέτες και εκθέσεις μας ε, που βρίσκονται και στο πίσω μέρος αίθουσας ε, τεκμηριώνουμε ακριβώς το πώς φτάσαμε σε αυτά τα νούμερα. Και έχω και κάποιες ερωτήσεις προς τους καλεσμένους σας. Καταρχήν, για να εξασφαλιστεί ο ανθρωπιστικό πυρήνα τη επανεγκατάσταση, θα πρέπει να δοθεί ένα επίσημο ε, και τυπικό ρόλο και στου ανθρωπιστικέ οργανώσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο κατά τη θέσπιση του ενωσιακού πλαισίου, αλλά και το θέμα τη αιτήσια εφαρμογή και παρακολούθηση εφαρμογή αυτού του ευρωπαϊκού πλαισίου επανεγκατάσταση. Τι γνώμη λοιπόν έχουν οι εμπειρογνώμονε, πώ θα μπορούσε να εξασφαλιστεί αυτή η συμμετοχή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι κατεξοδότηση πράξη και τη σύνθεση τη ε, Επιτροπή ε, Υψηλού Επιπέδου για την Κατάσταση. Επίση, ποια είναι η άποψή σα ε, για την ένταξη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συντονίσει και να διευκολύνει την ένταξη των προσφύγων στην Ευρώπη. Εκεί τεράστια προσπάθεια θα πρέπει να γίνει επιπλέον ίσως θα πρέπει να έχουμε κάποια υποχρεωτικά μέτρα και σε φάση πρώτης αναχώρησης και μετά την άφηξη. πώς θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την ένταξη και να αξιολογήσουμε το βαθμό της ένταξης μέσω κάποιων δικτών. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, στα μέλη του πάνελ, με τη σειρά που μίλησε και προηγουμένως. Στο τέλος θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να αντλήσει κάποια συμπεράσματα και να δώσει και τις δικές της αλλά πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Παρουσέλ και θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω τους εμπειρογνώμονές μας να είναι στο πιο λακωνική γίνεται. Και ο καθένας απαντάει σε ερωτήσεις που θεωρεί ότι τον αφορούν. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι τέθηκε συγκεκριμένη ερώτηση προς εμένα. Ως προς την πρόταση δεν έχω σχόλιο, γιατί εγώ είμαι ορμόδιος ε, για την εκπόνηση της συγκριτικής μελέτης και όχι αρμόδιος για το σχολιασμό της πρότασης ε, του πλαίσιου επανεγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της επανεγκατάστασης και αν η πρόταση θα αυξήσει ή θα μειώσει την επανεγκατάσταση, σε ανταπόκριση τη προσφυγική κρίση, πολλέ χώρε προσπάθησαν να κλείσουν τα σύνορά του, να γίνουν πιο αυστηρέ σε θέματα ασύλου, να θεσπίσουν κάποια περιοριστικά μέτρα και φυσικά η επανεγκατάσταση θα μπορούσε να έχει διαφορετική λειτουργία, να μην παρέχει μόνο προστασία. Γιατί θα μπορούσε η επανεγκατάσταση να γίνει μέτρο ε, ίσως ε, φυσικασμού των συνειδήσεων. Μερικές χώρες ξεκίνησαν προγράμματα επανεγκατάστασης, αυτό είναι πολύ θετικό. Θα πρέπει όμως ε, οι αριθμοί να αυξηθούν, γιατί για πολλές χώρες είναι πολύ μικροί οι αριθμοί, πολύ ελάχιστα τα ποσοστά επανεγκατάστασης. Οπότε το πρόγραμμα δίνει και ένα πολιτικό μήνυμα ότι κάνουμε και κάτι θετικό. Δεν κλείνουμε μόνο τα σύνορά μα, αλλά έχουμε και κάποιε θετικέ ενέργειε. Αλλά στο μέλλον θα πρέπει να προσέξουμε και του αριθμού. δεν θα πρέπει να μείνουν στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. Σα ευχαριστώ ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας ε, του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω συντομία να απαντήσω σε ό,τι αφορά το σύστημα των πόντων ε, για τις ευπάθειες. Εδώ μιλούσα, μιλήσαμε για την ταυτοποίηση των προσφύγων που χρειάζονται την επανεκατάσταση. Η διαδικασία ταυτοποίησης ξεκινάει από την καταχώρηση ενός πρόσφυγα στην υπετερμοστία, μετά γίνεται η επίσκεψη στην κοινότητα. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, δεν γίνεται για ένα για μια ενέργεια που γίνεται άπαξ και αποφασίζουμε όχι ε, πρόσφυγα ταυτοποιείται για την επανεγκατάσταση. Χρειάζεται γνώση για τον μεμονωμένο άνθρωπο, για τη συγκεκριμένη χώρα και πολλές γνώσεις σχετικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά του Σύρους, εκεί είχαμε εξαιρετικά στοιχεία για τους πρόσφυγες. Και τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά δεν, συγκεντρώνονται μόνο από την υπατερμοστή, αλλά από όλου του εταίρου μα, τι ανθρωπιστικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται σε γειτονικέ χώρε. Οπότε συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα δεδομένα σε μια πλατφόρμα που είναι προσιτή και σε εμά και με βάση αυτά τα στοιχεία βλέπουμε ποιοι συγκεκριμένοι πρόσφυγες έχουν μικρά παιδιά ή ε, αν έχει προηγηθεί κάποιο μέλος της οικογένειας ή σε ε, ποιους πυρήνες έχουμε ε, μόνη μητέρα. Γίνεται, γίνονται συνεχώς αυτέ ε, αυτές οι δραστηριότητες. Είναι μια δυναμική διαδικασία και είναι μοναδικός ο ρόλος της υπερσαρμοστίας. Ό,τι αφορά τη κοινωνικο-οικονομική ευπάθεια και το θέμα της οικογενειακής επανένωσης. Ό,τι αφορά την κοινωνικο-οικονομική ευπάθεια θα πρέπει να το ορίσουμε. Μερικοί επισημάνατε ότι πολλοί πρόσφυγες ε, θα ενέπταν ε, σε αυτό τον ορισμό, σε αυτό το χαρακτηριστικό. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε νέα κριτήρια επιλεξιμότητα. Τα υφιστάμενα συστήματα και για την υπατερμοστία και για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και για τα κράτη επανεγκατάσταση ε, εφαρμόστηκαν. Ε, ε, εφαρμόστηκαν τα υφιστάμενα κριτήρια. Τώρα με την καινοτομία και με την εφαρμογή νέων κριτηρίων που δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα, ίσως υπονομεύσουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος που είναι σημαντικές. Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή επανένωση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, γιατί η επέτερμοσία έχει ε, την την οικογενειακή επανένωση ως ένα από τα κριτήρια της επανεγκατάστασης. Για άτομα όμως που δεν μπορούν να βρουν άλλο νόμιμο, μια άλλη νόμιμη δίωδο και έχουν ως μόνη διέξοδο την οικογενειακή πανένωση. Τώρα να το θεωρήσουμε ως γενική προσέγγιση, οριζόντια, αυτό είναι σαν να μπερδεύουμε την οικογενειακή επανένωση με την επανεγκατάσταση. Γιατί οι ευκαιρίε επανεγκατάσταση είναι τόσο πολύτιμε, τόσο λίγε, τόσο ανεκτήμητε. Ε, είναι κρίμα λοιπόν να αφαιρούμε από την επανεγκατάσταση κάποιε θέσει και να ενισχύουμε την οικογενειακή επανένωση προσοχή να μην γίνει σύγχυση. Και τώρα, για την ερώτηση αν θα αυξηθούν οι αριθμοί τη επανεγκατάσταση. Αν θέλουμε να αυξηθούν τα ποσοστά επανεγκατάσταση, θα πρέπει η επανεγκατάσταση να συμπληρωθεί με άλλε νόμιμε διόδου και να μην τι υποκαθιστά. Και σίγουρα η οικογενειακή επανένωση είναι σημαντικό παράγοντα. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τα νούμερα, θα πρέπει ε, η επανεγκατάσταση να στηρίζεται στι ανάγκε, να είναι ε, μηχανισμός προστασίας ανθρωπιστικός, να έχει μια βιώσιμότητα, μια διάρκεια και φυσικά να εφοδιάζεται με τους απαραίτητους πόρους, ιδιαίτερα για την υποδοχή και την ένταξη. Αν λοιπόν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, τότε θα έχουμε πραγματικά και μεγαλύτερα ποσοστά επανεγκατάστασης. Μεταξύ του 2012 και του 2016, η αρμοστία του ΟΗΕ διπλασίασε τις ε, παραπομπές επανεγκατάστασης ε, από 700 σε 1500. Μέσα σε μία τετραετία διπλασιάστηκαν ε, οι παραπομπές, οι υποβολές. Μόνο σε μία διετία διπλασιάστηκαν και ήταν κέριο το σημείο, κρίσιμη στιγμή μετά τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης που είχαμε αύξηση διπλασιασμό των προτάσεων επανεγκατάστασης είναι σημαντικό το πρόγραμμα, θα πρέπει να στηρίζει τις ανάγκες, να αξιοποιεί υφιστάμενα πλαίσια. Έχουμε άλλους τρει ομιλητέ παρακαλώ, μην απεκτείνεστε. Πρέπει να προχωρήσουμε γιατί δεν ε, έχουμε χρόνο. Ναι, θα σταματήσω εδώ. Η Πέτρα για δύο-τρία λεπτά μόνο. Και πάλι όσον αφορά ε, τους αριθμούς, γιατί ε, με αυτό ασχολούμαστε και εδώ και 10 χρόνια προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς ε, μπορεί να εφαρμοστεί. Αν δείτε την εμπειρία των ε, σύρων ε, και τη δουλειά που κάνει η πατιαρμοστία, εξετάζει ξεχωριστά επιπλέον νόμιμες οδούς για την επανεκατάσταση. Πρόκειται για κάτι το οποίο ήταν επιτυχής. Εγώ ασχολήθηκα με πάνω από 130.000 θέσεις τότε. Ό,τι βλέπουμε τώρα σε αυτό τον κανονισμό είναι ότι τα πάντα συγχωνεύονται. η επανένωση των οικογενειών γίνεται τμήμα της επανεγκατάστασης, επομένως ο διαχωρισμός ε, των άλλων νόμιμων οδών σε σχέση με την επανεγκατάσταση ε, Συγχαίεται. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να έχουμε επιπλέον νόμιμους νόμιμες οδούς και επιπλέον στοιχεία. Επιπλέον αριθμούς ε, ανθρώπων μπορούμε να τα επιτύχουμε με άλλους τρόπους, με χορηγίες, αλλά μην το λέτε επανεγκατάσταση τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Όσκαρ Έκπλαν, παρακαλώ. Πολύ σύντομα για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την επανεγκατάσταση στην Ευρώπη και πώς μπορεί να γίνει. Από καθαρά διαχειριστικούς τρόπους, χωρίς να δούμε τι ικανότητα έχουμε απορρόφησης κλπ διότι αυτό μπορεί να είναι και πολιτική συζήτηση. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Οι Καναδοί έφτασαν στις 25.000 και πρόσθεσαν κι άλλες 10.000 μέσα σε λίγες ε, μήνες. Είναι εντυπωσιακό βέβαια αυτό, δεν θα το ξανακάνουν μάλλον από ό,τι ακούω, γιατί δεν γίνεται έτσι επανεγκατάσταση. Η επανεγκατάσταση είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση που πρέπει να προχωρήσει κλιμακωτά. Ε, δεν ε, ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση επανεγκατάσταση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε και τα διάφορα δομικά στοιχεία. την διαδικασία της είπα ένα καλό σύστημα υποδοχής εν τέλει που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Αν αυξηθεί σταδιακά και φτάσουμε σε αυτό, τότε η Ευρώπη έχει περιθώριο για να μπορέσει να καλύψει τα θέματα αυτά από πλευράς διαχείρισης. Ε, όσον αφορά ε, το, την ετοιμότητά μας. Εμείς γι' αυτό ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα από αυτού, για να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας. Ε, πέραν από τα πολιτικά στοιχεία, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και κάποια πρακτικά στοιχεία. Αυτό μαθαίνεται στην πράξη και όταν τα καταφέρουμε, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με βάση αυτό. Και τέλος, ο Πατρίς Κεσάδα από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Όπως ακούσατε υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκληση απόψεων ε, στο πάνελ. Μάλιστα υπάρχει πιθανότητα για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να προσθεθεί στα εθνικά προγράμματα που μπορεί να υποστηριχθεί από την Κομισιόν. Αλλά σε ένα βαθμό ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες σε τέτοιες προτάσεις ε, πρέπει να υπάρξουν κάποια πράγματα που θα ξεκαθαρίσουν στον κανονισμό με πληθυσμούς τόσο ευπαθείς, ε, ίσως να έχετε συναντήσει κάποιους, ε, δεν θέμα να είναι ανεπιτυχής η διαδικασία επαναγκατάστασης. Είναι πολύ μεγάλη επένδυση, οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση δύσκολη ε, οπότε, ναι, υπάρχει η πιθανότητα για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο σταδιακά θα αυξάνεται και θα οδηγήσει και θα πρέπει να έχει και μια ιδιαίτερη πτυχή ένταξης. Ναι, εσείς την ένταξη περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Τώρα θα ακούσουμε την εισηγήτριά μας. Μάλλον. Ε, απαντήστε στις ερωτήσεις, αλλά πείτε μας και τα συμπεράσματά σας και την προσέγγισή σας σε αυτή την έκθεση, που ξέρω ότι είναι δύσκολη όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν, οπότε πείτε μας ποια θα είναι η δικιά σας προσέγγιση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και το πάνελ και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που ήρθαν. Είναι δύσκολο το θέμα, όπως είπατε, γιατί υπάρχει, υπάρχουν κάποια προβληματικά άρθρα που χρειάζονται βελτίωση οπωσδήποτε και είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικό το θέμα και πρέπει να το βελτιώσουμε. Ο τελευταίος ομιλητής επίσης είπε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη σύγκληση αλλά και αποκλήσεις. Θα ήθελα εγώ να αναφέρω κάποια πράγματα που σημείωσα. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η επαναγκατάσταση δεν θα πρέπει να γίνει ένα εργαλείο για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Αυτό το βλέπουμε όχι μόνο με αυτήν την πρόταση, αλλά το έχουμε δει και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αναπτυξιακή Βοήθεια όπου είναι πάντα υπό τον όρο της συνεργασίας για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Και πρέπει να κάνουμε κάποιες σημαντικές επιλογές ως Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Και όπως είπαν πολλοί ομιλητές, η επαναγκατάσταση πρέπει να παραμείνει με βάση τις ανάγκες των ατόμων να είναι ένα εργαλείο προστασίας και αλληλεγγύης. είναι κάτι το οποίο πρέπει και εμείς ως Κοινοβούλιο να βελτιώσουμε οπωσδήποτε. Επίσης, βλέπουμε πως με τα κριτήρια πλεξιμότητας υπάρχουν κάποια προβληματικά σημεία, κάποια σημεία που πρέπει να τα σκεφτούμε περισσότερο, κάποια πρέπει να διαγραφούν ή να καθοριστούν καλύτερα. να κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, τους εκτοπισμένους και υπάρχουν κάποια σημεία που οπωσδήποτε πρέπει να διακρίνουμε την οικογενειακή επανένωση γιατί ε, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθούν οι αριθμοί αν υπάρξει μια σύγχυση και η οικογενειακή επανένωση μετά πάει στην επαναγκατάσταση. Οπότε τα κριτήρια επίσης αποκλεισμού πρέπει να τα ξαναδούμε γιατί φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε από την αρχή της ατομικής προστασίας και δεν θα πρέπει να τιμωρείται κανείς επειδή προσπάθησε να μπει παράτυπα και αν κάποιος επίσης απορριφθεί από μια χώρα απορρίπτεται από όλα τα κράτη-μέλη κάτι το οποίο δεν έχει πάρα πολύ νόημα και είναι ίσως άδικο και είναι και διακριτική μεταχείριση. Πολύ αναφέρατε την ένταξη και εδώ πέρα πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση για να μπει στο πλαίσιο αυτό. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Έχω τις προτάσεις σας για ένα ζήτημα το οποίο θέσετε πράγματι. Η αριθμοί έχω καλούς και οδησηγητές, θέλουμε να αυξήσουμε τους αριθμούς και βλέπουμε πως η πρόταση ως έχει ε, δεν έχει αυτά τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή και πρέπει να θεωρηθεί ως συμπλήρωμα άλλων νομίμων διόδων και πρέπει να βρεθεί και μια οικονομική και οργανωτική δομή για να αυξηθούν οι αριθμοί. Επίσης χαίρομαι που ακούω ότι ναι, είναι μια πρόκληση επιμελητίας οπωσδήποτε, αλλά υπάρχουν τόσες καλές εμπειρίες. Όχι μόνο στη Σουηδία, σε όλες τις χώρες που αναφέρθηκαν, Το πρέπει νομίζω να εκεί να βασιστούμε και να αυξήσουμε τους αριθμούς. Και έρχομαι έτσι στο τελευταίο σημείο που θέλω να συνεργαστούμε μαζί σας στενά για να πετύχουμε την αρχιτεκτονική για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό, θα αυξάνει τους αριθμούς, αλλά ε, δεν θα έχει μια παράλληλη, αλλά μια συμπληρωματική δομή για να αναπτυχθούν αυτά τα προγράμματα μαζί. Δεν είναι μια πρόκληση, έχουμε ήδη κάποιες ιδέες επιτάπητος. Έχουμε και τη σχετική σύνοδο κορυφής της ΥΠΑ της του ΟΗΕ και πώς ακριβώς θα επεκτείνουμε την τριμερή συνεργασία που είναι η βάση για τα προγράμματα επαναγκατάστασης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ. για να μας ε, πείτε αυτά τα οποία έχετε και ό,τι δεν μας είπατε σήμερα ελάτε ε, σε επαφή μαζί μας ε, είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι σκιώδεις εισηγητές και θα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Μαλίν. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ήρθαν σήμερα και όχι μόνο σήμερα αλλά και γενικώ βεβαίω να ευχαριστήσουν αλλού τον ΜΚΟ και που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Όπως είπε η Μάλλον η πρόκληση είναι τεράστια. Όχι μόνο εδώ αλλά και αλλού όπου επενδύουμε χρόνο και χρήμα για να έχουμε τις δομές αυτές στο πλαίσιο του πακέτου ασύλου και μάλλον καλή επιτυχία με το φάκελο. Um, Σας ευχαριστώ που ήρθατε στη δημόσια ακρόαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ένα ακόμη σημείο στη σημερινή μέρη σε διάταξη. και ευχαριστώ για την υπομονή που δείξατε γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε λοιπόν το σημείο 4, απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22 Σεπτεμβρίου 2016, παρουσίαση από την Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα μας παρουσιάσει τις ε, συνεκδικαστήσεις υποθέσεις ε, C14 15 και C116 15. Ο κύριος Καϊόλα από την νομική υπηρεσία θα μας κάνει την παρουσίαση των δύο αποφάσεων. Έχετε το λόγο κύριε Καϊόλα, αν είμαστε όλοι έτοιμοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του τρίτου σώματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 27 Σεπτεμβρίου 2016 αφορά δύο συνεκδικαστήσεις υποθέσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά Συμβουλίου που ζητούσαν ε, ακυρώσει πολλών αποφάσεων σε σχέση με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει, αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων, ταξινόμηση οχημάτων και δακτυλοσκοπικά δεδομένα. Οι, οι αποφάσει αυτέ υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο σε εφαρμοστικέ ε, αποφάσει μετά την απόφαση 615 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Ε, γνωστή απόφαση ΠΡΟΥΜ. Η απόφαση ΠΡΟΥΜ, όπως ξέρετε, υιοθετήθηκε πριν τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα, με στόχο τη συμπερίληψη της ε, τη ουσία των αποφάσεων τη συνθήκη Απρούμ στο νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποφάση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 22 Σεπτεμβρίου αποτελούν πολλών προσφυγών ακύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου που συνιστούσαν εφαρμοστικά μέτρα που υιοθέτησε το Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρώην τρίτου πυλώνα για να αντιληφθούμε το νομικό υπόβαθρο αυτών των υποθέσεων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπέβαλε ε, το επιχείρημα του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου 36 των μεταβατικών διατάξεων για τις πράξεις που υιοθετούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνθήκης πριν τη θέση ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας ε, πρέπει να ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να διατηρούν μόνο την ουσία των δράσεων του πρώην τρίτου πυλώνα και κάποιων ειδικών αποτελεσμάτων αυτών των πράξεων, όπως την έλλειψη άμεσου αποτελέσματος. Επιπλέον και κατά τη θέση του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλου 36 δεν έχει ως συνέπεια την διατήρηση ενίσχυα οποιασδήποτε διαδικασίας λήψης απόφασης που δεν ε, ισχύει επί του παρόντος και που ε, ρητά ακυρώθηκαν με τη θέση σε ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας. Παρ' όλα αυτά, το ΔΕΚ αποφάσισε ότι με τη θέση σε ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας ε, δεν αποκλείονται αυτόματα τα εφαρμοστικά μέτρα με βάση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων που προβλεπόταν με βάση τον προηγούμενο τρίτο πυλώνα στο μέτρο που η, απόφαση, η διαδικασία λαμβάνεται σε μια απόφαση του Συμβουλίου πριν τη θέση της ισχύς της Συνθήκης Λισαβόνας. Τούτου λεχθέντος και για να διευκρινιστεί το γενικότερο πλαίσιο, το γενικότερο νομικό πλαίσιο της απόφασης ε, και ιδιαίτερα για τις δύο υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ζήτησε ε, δύο, έθεσε δύο επιχειρήματα για την τεκμηρίωση των προσφυγών ακύρωσης. Καταρχήν, ε, θεώρησε ε, εσφαλμένη ε, η ελληπή τη νομική βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου. Και το δεύτερο επιχείρημα αφορά κάποια διαδικαστικά στοιχεία. Το πρώτο νομικό επιχείρημα ήταν σωστό και οδήγησε σε ακύρωση τη απόφαση του Συμβουλίου με βάση αυτό το επιχείρημα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν σκόπιμο για το λόγο αυτό να εξετάσει και το δεύτερο νομικό επιχείρημα. Με βάση το πρώτο ουσιαστικό επιχείρημα το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι όπω επιχειρηματολόγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η διαδικασία με βάση την οποία υιοθετήθηκαν οι δύο αφισβητούμενε διαδικασίε, δηλαδή το άρθρο 25 παράγραφο 2 τη ε, απόφαση ΠΡΟΥΜ ε, ήταν ασφαλμένε γιατί προβλέπουν εντελεχείς κανόνες για την υιοθέτηση μέτρων, όπως αυτά που μάλιστα μέτρων που είναι πιο περιοριστικά. Γιατί προβλέπουν ομοφωνία αντί για ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Σε σύγκριση με την διαδικασία που προβλέπεται από τις συνθήκες για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, έδωσε τη γνώμη του όπως ε, θα όφιλε με βάση τη διαδικασία για την ε, υιοθέτηση εφαρμοστικών μέτρων δυνάμει του τρίτου πυλώνα. Επίσης τονίζεται ότι το δικαστήριο αναφέρεται σε διατάξεις του τρίτου πυλώνα που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας κάτι που συνιστά μια πολύ διάζουσα κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το δικαστήριο έκρινε ότι με βάση τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 της απόφασης ΠΡΟΥΜ, το Συμβούλιο ε, παραβίασε τους κανόνες που προέβλεπε ο τρίτος πυλώνας και ως εκ τούτου παράνομα υιοθέτησε τις αφισβητούμενες αποφάσεις απαιτώντα μία ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και μάλιστα χωρί προηγούμενη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ω εκ τούτου, το δικαστήριο ε, κύρωσε τι αφισβητούμενε ε, αποφάσει όπω ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση τις ε, διαδικασίες που συμφώνησαν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει τα αποτελέσματα των αφισβητούμενων δράσεων μέχρι ότου θεσπιστούν οι νέε πράξεις που θα αντικαταστήσουν τις προηγούμενες και που θα πρέπει να αποφασιστούν να ληφθούν από το Συμβούλιο με βάση την ισχύουσα διαδικασία και άρα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και με άλλες έξι υποθέσεις, ε, με προσφυγές που ασκήσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του Συμβουλίου και με βάση τις οποίες ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καϊόλα. Ελπίζω... Δεν ξέρω αν κάποιος έθελε το λόγο. Κύριε Χαλάχο, γι' αυτό ήρθατε. Ήλπιζα ότι γι' αυτό είχατε έρθει. Κυρία Σίπελ, εσείς σίγουρα δεν ήρθατε γι' αυτό. Έχετε έρθει για τους συντονιστές. Κύριε Καϊόλα, όλες αυτές οι προσπάθειες ελπίζω να τις εκτίμησε κάποιος στο web stream. Τις εκτίμησα εγώ σίγουρα, να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ενημέρωση και τη γνωμοδότησή σας. Την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Έτσι ε, έχουμε και μια ανταμοιβή, ένα σύντομο διάλειμμα 10 λεπτών πριν από τους συντονιστές. Ευχαριστούμε κύριε Καϊόλα. 10 λεπτά διάλειμμα πριν από τη συνεδρία των συντονιστών. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, δεν πρέπει να βρίσκεται στους συντονιστές, ε, να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση είναι και κλεισμένα των θερών. Θα συνεχίσουμε στις 5.30. Ευχαριστώ και ελπίζω να άξιζε τον κόπο, κύριε Χαλάχου.